Okay, uh, dear colleagues, I think we could get started. Uh, συνάδελφοι, ξεκινήσουμε. Θα δούμε αν έρθει και κανείς. Πόσα άλλα μέλη της Επιτροπής θα έρθουν κατά την διάρκεια της ε, παρουσίασης. Ε, το Εργαστήριο Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις, Επιτέσματα και Προκλήσεις οργανώθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής μας για να προετοιμάσουμε την ακρόαση της νέας υποψήφιας επιτρόπου. Έχει χωριστεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος μιλάμε για τους διεθνείς οργανισμούς, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και τον ΟΣΑ που παρουσιάζουν τις στρατηγικές τους στο δεύτερο μέρος οι ειδικοί αναλύουν συγκεκριμένα πεδία πολιτικής ε, κατά τη διάρκεια ζωής ε, τους ε, σε σχέση με τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις τους. Όλες οι παρουσιάσεις είναι επίσης διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα μας. Και βεβαίως βρίσκονται μαζί με τα άλλα σχετικά έγγραφα. Ξεκινάμε λοιπόν με τους διεθνείς οργανισμούς και τον κύριο Χάιντς Κόλλερ, βοηθός Γενικός Διευθυντής και Περιφερειακός Διευθυντής για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας κύρια Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε για να παρουσιάσουμε την απόψή μας για το μέλλον της εργασίας σε μια επίκαιρη στιγμή και για τον οργανισμό μας που γιορτάζει την επαιτειό τους, αλλά και με τη νέα σύσταση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να πω πως έχουμε μια μακρόχρονη συνεργασία με τον συνάδελφο εδώ πέρα και τον ΩΣΑ δηλαδή. Ίσως ε, αρκετοί να μην γνωρίζετε πως το Διεθνές Γραφείο Εργασίας είναι το παλαιότερος οργανισμός στο σύστημα του ΟΗΕ. Δημιουργήθηκε το 1919 μετά από τον Μεγάλο Πόλεμο και την Επανάσταση του 1917. Είναι ο μόνος πολυμερής οργανισμός ε, και με τα τρία μέρη, κράτος, εργαζόμενους ε, και εργοδότες, ε, από 187 χώρες. Κάποια ορόσημα από την ιστορία μας. Το 1919 στο κεφάλαιο 30 της συνθήκης του Riverside υπήρχε σχετική πρόβλεψη για την κοινωνική δικαιοσύνη. 1944 η ε, διακήρυξη της Φιλαδέλφειας ότι η εργασία δεν είναι εμπόρευμα. 1959 το βραβείο Ειρήνης Νόμπελ, 2008 η σχετική ατζέντα και 2019 γιορτάζουμε την εκατοστή επέτειό μας με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση προς το μέλλον της ε, δουλειάς μας. Φανταστείτε δηλαδή έναν κόσμο χωρίς τον οργανισμό μας, χωρίς οχτάωρο χωρί Σαββατοκύριακα, χωρίς βασικό μισθό και κοινωνική προστασία. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια η εργατική νομοθεσία, ε, συνολικά 190 εργατικές συμβάσεις, έχει επηρεάσει την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο. Η ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάρα πολλά κοινά. Πολλές από τις ιδρυτικές αρχές του οργανισμού μας είναι και στις ρίζες ευρωπαϊκού... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ιστορικούς λόγους, ο ILO πάντα ε, είχε κινηθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έχουμε συνεργασία με όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με την Κομισιόν και με τα κράτη-μέλη που είναι οι μεγαλύτεροι δωρητές ε, στον οργανισμό μας. Έχουμε τακτικές διαβουλεύσεις με την Κομισιόν, με το Κοινοβούλιο και δημοσιεύσεις ε, για τον κοινωνικό πυλώνα, παραδείγματος χάρη κτλ. παίζει ένα σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κύρωση των συμβάσεων του ILO εσωτερικά γιατί όλα τα κράτη-μέλη είναι και κράτη-μέλη του ILO οπότε όλες οι συμβάσεις του ILO κυρώνονται από τα κράτη-μέλη και εξωτερικά προωθώντας ε, τις βασικές αυτές προδιαγραφές μέσω των εμπορικών ε, συμφωνιών και της αναπτυξιακής συνεργασίας. Σύντομα, για την εκατοστή επέτειό μας και την σχετική δήλωση, Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, κάποιες κινητήριες δυνάμεις αλλαγής στην παγκοσμιοποίηση, το περιβάλλον, η τεχνολογία, η δημογραφία. Ναι, ναι, α, μου είπαν ότι μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τα τελευταία 5-6 χρόνια ακολουθούμε την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω για το μέλλον της εργασίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε συμβουλευτεί και τα τρία μέρη ε, ανά τον κόσμο για το πώς φαντάζονται ότι θα είναι το μέλλον της εργασίας. Αυτό κατέληξε σε μία έκθεση παγκόσμια τον Ιανουάριο φέτος που παρουσιάζει το όραμα μας για έναν κόσμο με, έναν, ε, με ένα λαμπρότερο μέλλον. Τελικά λοιπόν είχαμε την διάσκεψή μας τον Ιούνιο του 2019 με πάνω από 6.000 αντιπροσώπους από 187 χώρες, 34 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και 137 υπουργού εργασίας που υιοθέτησαν την διακήρυξη των 100 ετών για το μέλλον της εργασίας και στο εθνικό επίπεδο και στην Παγκόσμια Επιτροπή και επιβεβαίωσε την άποψη ότι χρειαζόμαστε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για το μέλλον της δουλειάς. Για να το πω απλά, να μιλάμε για ανθρώπους, ε, για ψηφιοποίηση, για τεχνητή νοημοσύνη, ε, θα ακούσουν, αλλά θέλουν να μάθουν τι σημαίνει αυτό για μένα. Κινδυνεύει η δουλειά μου, χρειαζόμαστε νέες δεξιότητες, ποιος μπορεί να με βοηθήσει τα λοιπά. Οπότε, ειλικρινά, ο οργανισμός μας προσπαθεί ακριβώς να δει αυτήν την κοινωνική διάσταση του μέλλοντος της εργασίας. Η διακήρυξη αυτή έχει τρεις βασικές συστάσεις. Πρώτον, την ενίσχυση, και αυτό είναι σημαντικό, την επένδυση στις ε, δυνατότητες όλων των ανθρώπων για να ωφεληθούν από τις ευκαιρίες ε, του κόσμου της εργασίας ο οποίος αλλάζει μέσω και της ισότητας των φύλων αποτελεσματική διαβίου μάθηση παγκόσμια ε, κοινωνική προστασία και στήριξη στην μετάβαση στην, ε, στον εργασιακό βίο των ανθρώπων. Δεύτερον, ενίσχυση των θεσμών της εργασίας ε, μέσω της συμμόρφωσης ε, με το, τις βασικές συμβάσεις του ILO που λέγονται επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα στη δουλειά. Δηλαδή, ελευθερία του συνεταιρίζεστε και συλλογικές διαπραγματεύσεις, όχι καταναγκαστική εργασία, όχι παιδική εργασία και όχι διακρίσεις. Αλλά επίσης θέλουμε να δούμε και επαρκείς μισθούς ε, μέγιστο ωράριο και εγγυήσει για την ασφάλεια και την υγιεινή συνεργασία. Η δουλειά ε, δεν ε, θα πρέπει να σε ακροτηριάζει, να σε σκοτώνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τρίτη προτεραιότητα, προώθηση της βιώσιμης ε, ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και αξιοπρεπής αξιοπρεπούς εργασίας για όλους όπως αναφέρει και η ατζέντα του ΟΗΕ και συγκεκριμένα αναπτυξιακή στόχη. Ε, των οποίων ε, ο ΑΕΛΟ είναι θεματοφύλαξη εδώ πέρα, θα πρέπει να δούμε από πού προέρχονται οι δουλειέ του μέλλοντος. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στην ψηφιοποίηση, αλλά και σε κλασικούς ε, κλάδου. όπως η φροντίδα ανθρώπων και η δίκαιη μετάβαση στις πράσινες δουλειές. Όσον αφορά τώρα την συνοχή, αναμένουμε την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθήσει την ε, δήλωση της εκατοντατηρίδας που θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου. Ελπίζουμε να μην ενισχύσει μόνο την συνοχή μεταξύ μας, αλλά να δώσει και περαιτέρω κατευθύνσεις στους νέους επιτρόπους και τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να κινητοποιηθούν σε ζητήματα για το μέλλον της εργασία Τώρα, η σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της δουλειά. Πράγματι, κάνουμε μια κοινή διαδρομή για να διαμορφώσουμε το μέλλον της δουλειά, όπως το θέλουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε καλή θέση αν συνδυάσουμε την δήλωση του ΑΕΛΟ με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και τις προτάσεις ε, που έχει κάνει η ε, νέα πρόεδρος ε, της Κομισιόν και στο πρόγραμμά της και στις επιστολές που όπως ξέρετε βεβαίως θα τα εξετάσει όλα αυτά το Κοινοβούλιο της Ακροάσης. Καλωσορίζουμε ιδιαιτέρως το βάρος που δίνεται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ήμασταν παρόντες ε, τότε στη σύνοδο του Γκέντεμποργκ με τον γενικό μας διευθυντή γιατί ήθελε ακριβώς να διευθυνθεί την σύγκληση προς τα πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον κοινωνικό πυλώνα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο για να διαμορφώσει ένα δίκαιο μέλλον για την εργασία που θα επιλέγεται ελεύθερα και θα είναι αξιοπρεπής για όλους. Βλέπουμε ήδη πως ο πυλώνας έχει επιτύχει αυτά αποτελέσματα. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαιτέρως την οδηγία που ενεκρίθη πρόσφατα για την ε, ισορροπία ζωής και εργασίας για τους γονείς και όσους φροντίζουν τους δικούς τους. Αν μιλήσω στους νέους που έρχονται και ζητάνε δουλειά. Εμένα ζητούσα όταν ήμουν νέος προοπτικές, ίσως μία κάρτα κτλ. Σήμερα με ρωτάνε οι νέοι τι ευέλικτο ωράριο έχετε, τι μπορείτε να κάνετε για την ισορροπία ζωής και εργασίας. Αυτό έχει σημασία για τους νέους και πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Επίσης, ως κομμάτι της περαιτέρω εφαρμογής της αρχής της ισότητας των φύλων, μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το φύλλο που προβλέπει διαφάνεια στις ε, πληρωμές, στις διευθυντικές ε, θέσεις των εταιριών. Θα ταιριάξει πάρα πολύ καλά με την δήλωσή μας για τα 100 χρόνια του οργανισμού μας. Καλωσορίζουμε επίσης ε, την δέσμευση για την προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή και θα ήθελα τώρα να τονίσω δύο εκρεμή ζητήματα. Πρώτον, η δημιουργία ενός νέου νομικού μέσου για να διασφαλίσουμε ότι κάθε δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει έναν δίκαιο βασικό μισθό, κάτι το είναι ρεαλιστικό πλέον κατά την άποψή μας. Αυτό θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα στις δουλειέ των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επίσης ε, είναι και αυτό το οποίο ζήτησαν πολλές χώρες στην Γενέβη τον Ιούνιο στην δήλωσή μας η οποία σωστά αναφέρει ότι χρειάζεται ένας επαρκής βασικός ε, μισθός ε, είτε νομοθετημένος είτε που θα προκύπτει από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, θεωρούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ανεξαρτήτως από τον τύπο και διάρκεια της απασχόλησής τους, ε, θα συνεχίσουν να έχουν δικαίωμα σε επαρκή κοινωνική προστασία. Η συστάσεις ε, του Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου 2018 για την πρόσβαση στη, στα βοηθήματα από τους αυτοαποσχολούμενους είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Επίσης, να φροντίσουμε τα συστήματα κοινωνικής ε, προστασίας να ενισχυθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. και αυτό είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Επίσης, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τον σχεδιασμό ε, ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος αντασφάλισης επιδομάτων ανοιγίας. Ξέρω ότι είναι πολιτικά επίμαχο το ζήτημα. Και ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την κοινωνική προστασία για όλους και για τις νέες μορφές εργασίας και τις ε, μη συνηθισμένες μορφές εργασίας. Το Green New Deal το θέμα του κλίματος και του περιβάλλοντος ήδη επηρεάζει πολύ τον κόσμο της εργασίας. Σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε διεξάγεται στη Νέα Υόρκη η Σύνοδος Κορφής του ΕΕ για το κλίμα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο να δούμε ένα ευρωπαϊκό Green Deal και να υπάρξει μια δίκαιη μετάβαση για αυτούς που επηρεάζονται περισσότερο όπως τόνισε και η νέα πρόεδρος έτσι ώστε κανείς να μην μείνει πίσω. Κάτι το οποίο βεβαίως περιέχεται και στην ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030. Θεωρούμε πως υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας όπως δείχνει και η έρευνά μας. Εκτιμούμε στην Ευρώπη ένα καθαρό όφελος 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από μια μετάβαση προς την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Παγκοσμίω Μιλάμε για ένα κέρδος 18 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, όμως θα χαθούν ε, και δουλειές και αυτό είναι γεγονός. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη μετάβαση, έτσι ώστε οι προσπάθειες να προωθηθεί η πράσινη οικονομία θα πρέπει να συνοδευτούν από πολιτικές που θα προωθούν την ανακατανομή εργαζομένων, την επανεκπαιδευσή τους και καινοτόμα μέτρα κοινωνικής προστασίας. Δεν θα πρέπει να μείνουν ξεκρέμαστοι γενικά μιλώντας. Η πρωτοβουλία κλιματικής δράσης για τις δουλειές ενθαρρύνει τις χώρες να καταδίσουν σχετικά σχέδια μετάβασης. Επίσης θεωρούμε ότι όλα τα μέτρα αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε έναν κοινωνικό διάλογο ο οποίος θα λειτουργεί σωστά και ε, θα ε, παρέχει κοινωνική προστασία στους ευάλωτους. Ψηφιακή ατζέντα οι τεχνολογικέ εξελίξεις και συγκεκριμένα η ψηφιοποίηση επηρεάζουν πάρα πολύ τον κόσμο της δουλειά και τι εργασιακέ σχέσεις. Υπάρχουν ε, εδώ πέρα διάφορα πράγματα που μπορεί να κάνει ο ΑΕΛΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά όσον αφορά την ε, νομοθεσία, την εργασιακή, κατά το οποίο σας ενδιαφέρει προφανώς, και επενδύοντας ε, και πάλι στην εκπαίδευση και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων είναι δικαίως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το να κοιτάει και το τι μπορεί να γίνει με τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες συνολικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφής σχέση μεταξύ της ψηφιακής ατζέντα, της δίκαιης μετάβασης σε πράσινες δουλειές και της ατζέντα για τις δεξιότητες. Και η Επιτροπή μας ζήτησε την ε, σύσταση ενός, συστήματο ενός συστήματος διαβίου εκπαίδευσης και του δικαιώματος στην διαβίου εκπαίδευση. Και η διακήρυξη για τα 100 χρόνια ζητάει να προωθηθούν οι δεξιότητες και τα προσόντα για όλους τους εργαζόμενους ως κοινή ευθύνη κυβερνήσεων και κοινωνικών εταίρων. Σαφώς υπάρχει ανάγκη για καινοτόμες λύσεις με βάση τις κοινέ ευθύνες εργαζομένων, εργοδοτών και κυβερνήσεων όμως και αυτό είναι κάπως λύπηρο λίγες χώρες έχουν αναπτύξει ένα πλήρες πλαίσιο και καμία χώρα δεν έχει δημιουργήσει ένα σύστημα χρηματοδότησής του. Βεβαίως, ο κοινωνικός πυλώνας ε, περιέχει το δικαίωμα ποιοτική κατάρτισης για όλους, οπότε θα μπορούσε να υπάρξει μια εγγύηση διαβίου κατάρτισης ε, μαζί με την εγγύηση για την νεολαία για τα άτομα 125. Οπωσδήποτε ένα σημαντικό ζήτημα είναι η δημιουργία λογαριασμών μάθησης για τους ε, νέους ε, και τους εργαζόμενους. Τέλος, αναφέρατε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Παρακολουθούσαμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον την φιλοδοξία της νέας Προέδρου να αποτελέσει μια γεωπολιτική κομισιόν. Αυτό Βεβαίω, ε, μας συγκινεί ως ε, διεθνή οργανισμό και πολύ περισσότερο μας αρέσει το ότι ο κάθε επίτροπος καλείται να ενσωματώσει την ατζέντα των αναπτυξιακών στόχων στο χαρτοφυλάκιο του. Αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική βελτίωση. Δύο λόγια τώρα για τους κοινωνικούς εταίρους. Ακόμα και στην Ευρώπη είχαμε μια επιδύναμη, επιδύνωση των συλλογικών ε, διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου. Όχι μόνο λόγω της οικονομικής χρήσης, αλλά και το αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της απορρίθμισης. Αναφέρομαι στον ΟΣΑ. Οι χώρες ΟΣΑ Εκεί 30% των εργατών ήταν μέλη συνδικάτων το 85% και μόνο 17% σήμερα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αναζωογονήσουμε τον κοινωνικό διάλογο. Κυρίως ε, όσον αφορά τις νέες μορφές εργασίας. Κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοπρεπής εργασία και ανθρωποκεντρική ατζέντα για τον 21ο αιώνα πρέπει να είναι κοινή μας στόχη. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο είναι στην πρώτη γραμμή και ελπίζουμε ότι και αυτό θα είναι κάτι που θα διδοθεί και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Τέλειος ο χρονισμός σας. Θα να ακούσω ερωτήσεις, συστάσεις. Οι συντονιστές, υπάρχει κάποιος από εσά ο οποίος επιθυμεί να θέσει ερώτηση. Όχι. Άλλα μέλη της Επιτροπής. Καλώς. Η παρουσίαση ήταν τέλεια. Δεν υπάρχουν καν ερωτήσεις. Πάμε στο θεματολόγιο της μετάβασης για το μέλλον, προς το μέλλον, δουλειές για όλους. Ο κ. Καρπέτα, Διευθυντής για Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις του ΟΣΑ, θα λάβει το λόγο να αναφερθεί στο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη της Επιτροπής, μεγάλη χαρά για μένα να συμμετέχω σε αυτό το εργαστήριο. Έτσι θα μοιραστώ κάποια βασικά σημεία των εργασιών του ΩΣΑΑ. Τα χρόνια αυτά να αξιολογήσουμε την ψηφιακή μετάβαση και πώς οι άλλες μεγάλες αλλαγές αλλάζουν την αγορά εργασίας και τις οικονομίες μας. Όταν μιλάμε για τη μελλοντική εργασία, όπως είπε και ο Χάιντς, αυτό είναι ένα θέμα που πολύ συχνά δημιουργεί ανησυχία. Βομβαρδιζόμαστε με πληροφορίες για δουλειές που θα εξαφανιστούν, για ένα μέλλον χωρίς εργασία, τα ρομπότ που θα μας επιβάλλουν πρέπει να κάνουν στη δουλειά μας κλπ. Σε αυτό το τομέα, όπως και σε άλλους, είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάσουμε τα στοιχεία και να δούμε πώς η πολιτική μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα, να προβλέψει τις αλλαγές και να ανοίξει ευκαιρίες που θα μας δώσει η ψηφιακή μετάβαση. Το πρώτο που έχω να πω, βασισμένο σε αυτά που είπε ο Χάινς, είναι το εξή. Αντιμετωπίζουμε τρεις μεγάλες τάσεις και όχι μία. Η ψηφιακή μεταμόρφωση αλλάζει τάχιστα και εις βάθος τις οικονομίες μας και τις αγορές εργασίας. Βλέπετε τέσσερις από τις δέκα θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες του ΟΣΑ είναι σε τομείς ε, που είναι εντατικά ψηφιοποιημένοι σε σχέση με το παρελθόν. Όταν δεξιά βλέπετε ότι οι οικονομίες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και στις περισσότερες χώρες του ΟΣΑ γυράσκουν τάχιστα οι πληθυσμοί μας. Ένα στους τέσσερις είναι από 65 και πάνω στους τέσσερις για τέσσερι, που είναι σε ηλικία εργασία το 2050 κατά μέσο όρο στι χώρε ΩΣΑ ένα στου δύο θα είναι πάνω από 65 και σε κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε η γύρανση θα είναι πιο γρήγορη 7 άτομα στα 10 θα είναι ηλικιωμένοι. Οι δημογραφικές αλλαγές αναδιαμορφώνουν και σε σημαντικό βαθμό τις οικονομίες μας και τις αγορές εργασίας μας. Και οι οικονομίες μας όλο και περισσότερο ολοκληρώνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπετε ότι πάνω από 40% των εργαζομένων στι χώρε ΩΣΑ και περίπου 50% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται για ξένους πελάτες, για ζήτηση σε άλλες χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ενώσης αλλά και εκτός αυτών. Οι οικονομίες μας είναι αλληλένδετες μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού και ολοκλήρωση σημαίνει ότι οι οικονομίες μας ε, έχουν αλληλεπίδραση. Αυτές είναι οι μεγάλες τάσεις λοιπόν που διαπιστώνουμε. Πρώτη ερώτηση εξ αυτών. Βλέπουμε ένα μέλλον χωρίς εργασία. Τι στοιχεία έχουμε. Τι παρατηρούμε από τα στοιχεία. Η απάντηση ουσιαστικά είναι ουχή. Αν δείτε τα ποσοστά απασχόληση, δηλαδή εκείνου που σε ηλικία εργασία έχουν δουλειά, στην Ευρώπη και στις περισσότερες χώρες ΩΣΑ είμαστε στα ύψιστα επίπεδα, ρεκόρ έχουμε πιάσει ε, κυρίως στη μεταποδομική περίοδο. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις χώρες. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, παρά κάποιες βελτιώσεις κατά παρελθόν, έχουν υψηλά επίπεδα ακόμα ανεργίας, αλλά ουσιαστικά η οικονομία μας όλο και περισσότερους ανθρώπους απορροφούν στις απασχόλησει, Όλο και περισσότερες ε, γυναίκες, αλλά και περισσότεροι εργαζόμενοι μένουν επί μακρύτερο χρονικό διάστημα στην απασχόληση. Δεν έχει μειωθεί ε, το επίπεδο απασχόλησης Παρ' όλα αυτά έχουμε αλλαγές τεχνολογικές. Περίπου το 1 τέταρτο τη μεταπίεση ε, έχει με, μεταπτικό τομέα έχει υποχωρήσει κατά 20%. Ενώ ο τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 22%. Δεν είναι οι ίδιε οι εργασίε, το είδο τη δουλειά, ο τόπο που γίνεται η δουλειά ε, και ε, ο τομέα που παράγει οι θέσει απασχόληση αλλάζουν σημαντικά. Ε, γιατί γίνονται αυτές οι συζητήσει για το μέλλον και τον κίνδυνο να μην υπάρχουν θέσεις εργασίας. Η τεχνολογία είναι άκρως διζητική και γρήγορες αλλαγές. Βλέπετε στο διάγραμμα αριστερά, σε παγκόσμιο επίπεδο, την παροχή βιομηχανικών ρομπότ από λιγότερο από 100.000 μέσα του 2005 πάμε σε 500.000 το 2017 και η προβολή που βλέπετε μέχρι να φτάσουμε 700.000 το χρόνο ε, το 2021 βιομηχανικά ρομπότ. Εκθετική η αύξηση του αριθμού των βιομηχανικών ρομπότ που μπαίνουν στην παραγωγή. Τι είναι το ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο αριθμό των ρομπότ, αλλά και ένα άλλο γεγονό ότι να έχει κανεί ένα ρομπότ και το χρησιμοποιεί στην παραγωγή κοστίζει στη ΣΥΠΑ ανάμεσα στα 10 και 20 δολάρια την ώρα. Σχεδόν λιγότερα από αυτό που κοστίζει ένα εργάτη στην παραγωγή. Οπότε αλλάζει η παραγωγή πολύ γρήγορα. Αν προβάλλουμε τι γίνεται στο μέλλον. Να πω σαφώ ότι υπάρχουν τεράστιε αβεβαιότητε για το μέλλον και πώ θα μπει στην παραγωγή τεχνολογία. Κάναμε μια εκτιμήσει στον ΩΣΑ πόσε θέσει απασχόληση κινδυνεύουν ή ενδεχομένω θα αυτομετωπιθούν. Τι σημαίνει αυτό. Ότι θέσει απασχόληση για το 70% περισσότερα από τα καθήκοντα γίνονται από εργαζομένου θα μπορούσαν να γίνουν από αλγόριθμο, τεχνητή νοημοσύνη ή κάποιο μηχάνημα Κάποια από τα στοιχεία που κυκλοφορούν και στα ΜΜΕ και λοιπά και στο μέσα κινητική δικτύωση έλεγαν ότι περίπου μισέ από τι θέσει απασχόληση θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν. Κατά τι εκτιμήσει μα, εμεί λέμε ότι είναι περίπου 14% κατά μέσο όρο στον ΩΣΑ και άντε 17% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ λιγότερο από αυτά τα αποκαλυπτικά στοιχεία που μας λένε για το μέλλον εκεί που τα περισσότερα καθήκοντα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από μηχανήματα. Δείτε όμως το διάγραμμα κάτω, υπάρχει ένα άλλο 32%, καμία φορά περισσότερο, ο οποίο παραμείνει η θέση απασχόληση, αλλά εφή τη δουλειά να αλλάξει σημαντικά, διότι σημαντικό ποσοστό των καθηκόντων που γίνονται στου εργάτε θα μπορούσαν να γίνουν από μηχάνημα. Ο εργάτη που έκατε στη θέση του, αλλά εκείνο ή θα πρέπει να προσαρμοστούν κάνοντα διαφορετικέ δουλειέ που θα συμπληρωματικέ από αυτέ που μπορεί να κάνει το μηχάνημα. Θα μπορούσε, λέω, λέω θα μπορούσε, διότι ο τρόπος με τον οποίο θετηθεί η νέα τεχνολογία εξαρτάται από την πολιτική, την επιλογή των εταιριών και την επιλογή της κοινωνίας. Δεν είναι ένα μέλλον χωρίς δουλειές, αλλά μέλλον όπου θα έχουμε βαθιές ε, μεταμορφώσεις και αλλαγές και όπου πολλές θέσεις θα δημιουργηθούν, απασχόλησεις ποιοτικέ με υψηλή αμοιβή και ενδεχόμενο δυνατότητα καριέρας αλλά και θέσεις που θα πληρώνουν λιγότερο και δεν θα είναι και τόσο καλές για την καριέρα κάποιου. Και ο Χάινς το είπε αυτό. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι πώς θα επιτρέψουμε στους εργαζομένους, όλους, όχι μόνο τους νέους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, όλους εκείνους που ήδη είναι στην αγορά εργασίας, να αποκτήσουν τι δεξιότητε που δώσουν δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν καλά στην εργασία του και να αποκτήσουν αυτέ τι δεξιότητε και γνώσει που θα είναι συμπληρωματικέ στο φάτι το τι μπορεί να κάνει η μηχανή. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Αριστερά βλέπετε πόσα άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά συμμετέχουν σε επίσημη και άτυπη κατάρτιση και βλέπετε ότι οι χαμηλέ δεξιότητε σε σχέση με αυτού που έχουν πολλέ δεξιότητε, αυτοί που κινδυνεύουν πολύ από τον αυτοματισμό σε σχέση που έχουν λιγότερο κίνδυνο. αυτοαποσχολούμενοι, προσωρινοί εργαζόμενοι, όλοι αυτοί είναι πιο ευάλωτε ομάδε και έχουν πολύ λιγότερη κατάρτιση από εκείνους που κινδυνεύουν λιγότερα από αυτοματοποίηση, αυτές που έχουν πολλές δεξιότητες που χρειάζονται λιγότερη κατάρτιση και ανα... επανεκπαίδευση. Είτε στη Σουηδία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία, στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά, όπου και να όλα τα συστήματα δίνουν περισσότερε περισσότερες δυνατότητε στι μεγάλε επιχειρήσει, αυτού που έχουν πολλέ γνώσει και δεξιότητε, και λιγότερε δυνατότητε εκείνου που κινδυνεύουν περισσότερο τον χρωματισμό και δεν έχουν πολλές δεξιότητες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεξιά βλέπετε ότι 6 στου 10 ενήλικες έχουν πολύ περιορισμένε ψηφιακέ δεξιότητε. Δεν λέω να, είναι, να κωδικοποιούν προγράμματα, δεν θα χρησιμοποιήσουν ψηφιακή τεχνολογία παραγωγικά στη θέση εργασία. Αυτό βέβαια είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι πάρα πολλέ από τι θέσει θα συμπεριλαμβάνουν και κάποιο στοιχείο ψηφιακών δεξιοτήτων. Ποιε είναι οι πολιτικέ που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν τι λέμε συστάσει πολιτική, διότι είναι ένα φάσμα δράσεων που μπορούν να εφαρμοσουν διαφορετικά Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να μπούμε είναι ότι πραγματικά θα πρέπει να μην αποφύγουμε ριζική επανάσταση, να θεωρήσουμε, όπως έλεγε ο Χάινς, ότι η διαβίω εκμάθηση είναι γεγονός. Όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες ε, κατά τη διάρκεια της ζωής τους στην εργασία. Ε, ε, να, τα εμπόδια για την κατάσταση να απομακρυνθούν και πρέπει οι εργοδότες να επενδύσουν και στου ανθρώπου με πολλέ δεξιότητε και λιγότερε και να δοθεί κάποια δημόσια υποστήριξη, να βοηθήσουμε και τι εταιρείε και του εργαζομένου να κατανοήσουν τι είδου κατάρτιση και τι είδου αρμοδιότητε και δεξιότητε χρειάζονται. Πρέπει τα δικαιώματα κατάρτιση να μπορούν να μεταφέρονται από δουλειά σε δουλειά δεν θα, πρέπει να, δεν θα κρατάει ένα την ίδια δουλειά σε όλη τη ζωή. Θα πρέπει ένα άτομο να μπορεί να έχει πολλέ καριέρε, πολλέ δουλειέ και πολλέ δουλειέ ταυτόχρονα ή πολλέ κατά τη ζωή του. Ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα εντόπισε ήδη κάποιε βασικέ αρχέ πολιτική και δράσει που θα μπορούσαν να δρομολογηθούν. Ωστόσο, σε κάποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με αυτό προχωράει, είναι προθυμένη και υπάρχουν κάποια διαφορετικά πειράματα όσον αφορά από την εκπαίδευση ατόμων ε, που αναφέρθηκε πριν και σε άλλε κατατάξει. Το εγγύηση για του νέου, το θεματολόγιο για τι δεξιότητε, η στάση του Συμβουλίου για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι μόνο κάποια μονοπάτια που υπάρχουν στο θεματολόγιο. Το δεύτερο σημείο που ίσω σα εκπλήσει, διότι στην Ευρώπη έχετε το σύστημα που έχει τη μεγαλύτερη κοινωνική προστασία. Αν δείτε όχι στα δικαιώματα και τι αξιώσει, αλλά την κάλυψη των ανθρώπων, θα δείτε ότι η αριθμή των εργαζομένων είναι μεγάλο που δεν καλύπτονται, ακόμα και έναντι του κινδύνου τη ανεργία. σω να καλύπτονται μόνο βραχυπρόθεσμα από την ανεργία. Σε όλε τι χώρε, ΟΣΑ και Ευρωπαϊκή Ενώση, δύο στου τρει ανθρώπου ε, που ψάχνουν για δουλειά δεν έχουν επίδομα ανεργία. Και αυτό είναι ιδιαίτερα πρόβλημα για εκείνου που ακολουθούν άτυπη μορφή εργασία. Δεν μιλάω μόνο για εργαζομένου κλασικά σε αυτού προσωρινού, ε, ε, συμβάσει ορισμένου χρόνου, αορίστου χρόνου κλπ που ίσως να βγάζουν λιγότερα από αυτούς που έχουν πιο τυπικές μορφές εργασίας. 40-50% από αυτούς που έχουν άτυπη μορφή απασχόλησης πιθανότατα δεν θα έχουν υποστήριξη στο εισόδημά του ε, όταν χάσουν. 40-50% λιγότερε πιθανότητε έχουν υποστήριξη στο σώδημά του όταν μείνουν άνεργοι. Ποιε κατευθύνσει προτείνουμε, Πρέπει να θεωρήσουμε την κοινωνική προστασία και τα δικαιώματα και τα κριτήρια να δώσουν πρόσβαση στην κοινωνική προστασία σε περισσότερου εργαζομένου σε άτυπη μορφή εργασία, δώσουμε τότε εργαζομένου σαν ανεκάτες μορφέ απασχόληση να δημιουργήσουν δικαιώματα για να υποστηριχτούν όταν έχουν δουλειά, να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε ε, τον επιμερισμό του κινδύνου στον αγορά εργασία και στα ομάδε εισοδημάτων, δίνοντα οικονομικά κινήτρα που ευνοούν άτυπε μορφέ εργασία, θα πρέπει να μεταφέρουν τα δικαιώματα σε διάφορε απασχόληση και μορφέ απασχόληση. Πρέπει να ενισχύσουμε καθολικέ ε, μορφέ υποστήριξη ανεφόρων και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη κάποια εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε τώρα πάνω σε αυτό. Τρίτον, και ίσω το σημαντικότερο σημείο είναι στην Ευρώπη και σε όλε τι χώρες του ΩΣΑ, η πρόσβαση στην προστασία των απασχολωμένων, στην κοινωνική προστασία, γίνεται μέσω τη σύμβαση, μέσω τη σύμβαση εργασία. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε λοιπόν τι συνθήκε που καθορίζουν ποιο είναι εργοδότη, ποιο είναι, αυτο... εργαζόμενο, ποιο είναι ανεξάρτητο εργαζόμενο και ποιο αυτοασχολούμενο. Ένα στου εννιά εργαζόμενου στι χώρε ΩΣΑ και ένα στου 7 στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προσωρινή σύμβαση ορισμένου χρόνου και όλοι μαζί άτυπε μορφέ εργασία είναι ένα τρίτο τη συνολική απασχόληση. Η σύμβαση απασχόληση είναι μια πύληση πρόσβαση προστασία κοινωνική και απασχόληση και γι' αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει σωστά να ταξινομούνται οι εργαζόμενοι ανάλογα με τη φύση τη δουλειά που κάνουν. Πράγματι, πράγματι, ένα στου 7 εργαζομένου στι χώρε του ΟΣΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοαπασχολούμενοι αλλά 16% των αυτοαποσχολούμενων οικονομικά εξαρτώνται από έναν πελάτη. Λοιπόν, κάποιο από του κράτου εργαζομένου μοιράζεται κάποια χαρακτηριστικά και τον ευαλωτότητα των εργαζομένων. σω να απολαμβάνουν κάποιο βαθμό αυτονομία, ίσω αποφασίζουν πού και πότε και πώ να εργαστούν, ίσω να εξαρτώνται όμω από έναν μοναδικό πελάτη για την παρεχόμενη υπηρεσία. Και γι' αυτό έχουν σημαντικό βαθμό εξάρτηση που ίσω του κάνει να είναι παρόμοιοι με τον εργαζόμενο, τον υπάλληλο. Ταξινόμηση των συμβάσεων και θα πρέπει να επιβάλλουμε και τους νόμους περιεργασίας. Λοιπόν, ποιε είναι από τι κατευθύνσει πολιτική από το τομέα να αντιμετωπίσουμε την ψεύτο αυτοαποσχόληση. Όταν το κάνουμε αυτό, πρέπει να ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που είναι στην κρίζα ζώνη. Δηλαδή, πράγματι, ίσω να έχουν κάποια επίπεδο ανεξαρτησία, από την άλλη πλευρά όμω, ίσω να, να είναι ανεξάρτητοι εργαζόμενοι και εξαρτώμενοι. Πρέπει να ξεκαθαρίζεται ποια είναι σχέση με τον εργοδότη και τον πελάτη και θα πρέπει να επεκταθεί η προστασία σε εκείνου που παραμένουν σε μια γκρίζα ζώνη. Η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία πρέπει να αυξηθεί, να επεκταθεί η πρόσβαση στην κατάρτιση, επανακατάρτιση και Λοιπόν, καταρχά να εξασφαλίσουμε ότι η ταξινόμηση είναι σωστή, ξεκάθαρη και να ασχοληθούμε με εκείνου που παραμένουν σε μια γκρίζα ζώνη. Εκεί είναι διάφοροι από εκείνου που είναι στη βασική οικονομία και εκείνου που ίσω να είναι όλο και περισσότερο στο μέλλον σε άλλε θέσει. Θα πρέπει να, να δούμε Ποιο ανήκει πού σε ποια κατηγορία. Και κάτι άλλο που επεξεργαζόμαστε στον ΩΣΑ. Σε κάποιου τομεί, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας εργαζόμενος που έχει ε, ε, μονοπόλιο σε έναν τομέα. Πρέπει Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζομένων. Έχει ένα είδους μονοπόλιο εργοδότης. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να πω κάτι που ανέφερε και ο Χάιν. Μιλάμε για τον εργαζόμενο που έχει μεγαλύτερο κίνδυνο που συνδέεται με τι οικονομίε μα Ταυτόχρονα και η αντιπροσώπευσή του μειώνεται. Κλασικό δείκτη. Βλέπετε, ότι με την πάγω του χρόνου η εντατικότητα τη εργασία μειώνεται. Σε κάποιου τομεί όμω ε, δεν καλύπτονται από συλλογικέ συμβάσει ή μορφέ εργασία. Όχι μόνο λιγότεροι εργαζόμενοι είναι μέλη ε, συνδικάτων, αλλά και εκεί που υπάρχουν συμφωνίε συλλογικέ και επεκτείνουν σε εργαζόμενου που δεν είναι μέλη των ενώσεων. Σε κάποιου τομεί ε, πολλοί εργαζόμενοι δεν καλύπτονται τι συλλογικέ συμβάσει. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εκπροσώπηση εργαζομένων, μεγαλύτερο κοινωνικό διάλογο σε μια στιγμή που παραδοσιακοί οι θεσμοί έχουν αποδυναμωθεί με την πάρα του χρόνου. Υπάρχουν κάποιε κατευθύνσει προσανατολισμού που τονίσαμε. Να συνοδεύσουμε την προσπάθεια των συνδικάτων και οργανώσεων εργοδοτών να επεκτείνουν τα αριθμό των μελών χωρί να αποθυράνουν την ε, ανάδυση νέων μορφών οργάνωση, να παρήσουμε περιθώριο για συλλογικέ συμβάσει και να δώσουμε κίνητρα για αυτορύθμιση μεταξύ των φορέων, ούτω ώστε να κάνουμε περιορισμένη στατική χρήση ε, νομοθετικών παρεμβάσεων, να προωθήσουμε εθνικέ διαβουλεύσει και συζητήσει για το μέλλον των εργασιών, τη εργασία. Σε αυτό το τομέα λοιπόν συμβαίνουν πολλά στην Ευρώπη, αλλά και σε όλε τι χώρε του ΩΣΑ. Κάποιε χώρε έχουν προωθήσει και προωθούν Νέε μορφέ οργανώσεω των εργαζομένων και σε κάποιο βαθμό υποστηρίζουν αυτέ τι νέε μορφέ οργάνωσης και κατά την άποψή μου αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να κλείσω αναφερόμενο σε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ που αφορούν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον αφορά τις πρέπει να αναζωογονήσουμε, επεκτείνουμε τι συλλογικέ συμβάσει και να αντιμετωπίσουμε την, τα μονοπόλια που έχουν κάποιοι εργοδότε. Αυτό πρέπει να το προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωπαϊκέ χώρε για του βασικού εργαζόμενου κλασικού πρέπει να τι και να την ταξινόμηση και τα δικαιώματα προστασία όσον αφορά των ευαλωτών αυτοαποσχολουμένων. Δεν λέμε να επεκτείνουμε την κοινωνική προστασία σε όλου του αυτοαποσχολουμένου. Κάποιοι από αυτοί έχουν επαρκά εισοδήματα και μπορούν να αυτασφαλιστούν. Αλλά για άλλου είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι έχουν την ίδια ευαλωτότητα με παραδοσιακού εργαζομένου. Κοινωνική προστασία πρέπει να ενισχύσουμε τα συστήματα κοινωνική προστασία, ώστε λιγότεροι άνθρωποι να πέφτουν σε κενά που υπάρχουν. Πολλέ σε, μία μη άτυπε μορφέ απασχόληση μπορούν να πέσουν μέσα σε κενά, ακόμα και σε πιο ανεπτυγμένα συστήματα κοινωνική προστασία που υπάρχουν στην Ευρώπη. Σαν τι δεξιότητε, νομίζω ότι είναι απόλυτα θεμελιώδε η διαβίω εκμάθηση να γίνει μια πραγματικότητα, αλλά αυτό δεν λειτουργεί ούτε καν σε χώρε που ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για να εκπαιδεύουν του ενήλικε. Δεν συμβαίνει για αυτού που το χρειάζονται περισσότερο και το τονίζω αυτό. Δεν λειτουργεί αυτού που έχουν χαμηλέ δεξιότητε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, δεν λειτουργεί για εκείνου που είναι μεσήλικες ή πιο ηλικημένοι. Εκείνοι που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα να κρατήσουν τη θέση απασχόληση και να μπουν στη δυναμική, πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό, ο κοινωνικός διάλογος, να επεκτείνουμε τη συλλογική διαπραγμάτευση σε κάποιε ομάδε αυτοπασχολουμένων εργαζομένων, να δημιουργήσουμε νέε μορφέ διαλόγου και κοινωνικού διαλόγου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Κλείνοντα, στα δύο λεπτά που έχω, να πω το εξή τελικά. Αυτά που είπα και αυτά που έλεγε και ο Χάιντς. Έχουμε μια ομάδα σημαντικών προβλημάτων αλλά και πολιτικών που ήδη οι χώρες θα πρέπει να δρομολογήσουν στο μέλλον. Δράση στο περιθώριο. Δηλαδή να διορθωθούν κάποια προβλήματα όσον αφορά τι ρυθμίσει για τα ενεργασία στην νομοθεσία, κοινωνική προστασία, για την κατάρτιση ξεχωριστά και αμή συνδέονται όλα μαζί, δεν θα γίνει. Θέλει ενιαία προσέγγιση. Το ILO και ο ΣΑ το λένε συχνά, αλλά μια ολιστική προσέγγιση χρειάζεται θα πρέπει όλα τα διάφορα στοιχεία να συναθριστούν, να συγκεραστούν και να δώσουμε μια πολιτική που θα δώσει απάντηση, ένα πακέτο που θα αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και να επιτρέψουμε και στου ανθρώπου να αρπάξουν τι προσφερόμενες ευκαιρίε. Διαβίω εκμάθηση δεν είναι μόνο θέμα πόρων, είναι ένα θέμα τη επαφή με του κοινωνικού εταίρου. Θα πρέπει ο κόσμο να γνωρίζει γιατί πρέπει να κατατεστεί και οι εργοδότε να έχουν τα σωστά κινήτα να εκπαιδεύσουν του εργαζομένου, όχι μόνο αυτού που έχουν ψηλέ δεξιότητε, με επαρκή χρηματοδότηση, δεν είναι μόνο ανακατανομή των πόρων στον ίδιο, στο κοινωνική, πολιτική, απασχόληση κλπ. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και πόρου από άλλα τμήματα τη κυβέρνηση, από άλλου κλάδου και αυτό είναι πάρα πολύ ένα θέμα θεματολογίου του ΟΣΑ. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλε οι επιχειρήσει να πληρώσουν του φόρου του. Το δίκαιο φόρο, όλοι θα γνωρίζετε, τα BEPS. Λοιπόν, είναι η πρωτοβουλία προωθεί ΣΑ όσον αφορά τα πλαίσια του G20, ότι όσοι πολυεθνικέ να πληρώνουν δίκαιους φόρους, να πληρώνουν τους φόρους βάσει των κερδών του. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία από τι πολλέ που εξασφαλίζουν ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει ο εταιρικό φόρο, αλλά όλοι θα πρέπει να πληρώσουν του φόρου, να μην ξεφεύγουν. Έτσι οι πόροι θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν προ μια θεματολόγια για τη μετάβαση τη οικονομία. Είναι ένα μεγάλο θέμα, φιλόδοξο πρόγραμμα που θα πρέπει να δρομολογηθεί τόσο ώστε να δώσουμε την απάντηση στον κόσμο εκείνων που ανησυχεί για το μέλλον τη εργασία. Και περιμένουν από όλου μα τι απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ακούσουμε τις δικές σας ερωτήσεις. Πρώτα οι συντονιστές. Ο κύριος Φίσλερ βλέπω. Θέλει να θέσει ερώτηση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή σας ε, την ε, παρουσίαση. Θέλω να υποβάλω στοχευμένες ερωτήσεις. Μήπως θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τις αδυναμίες και να μεταμορφώσουμε σε ε, δυνατότητες, να μετατρέψουμε την οικονομία και και έτσι να αναπτύξουμε μάλλον την οικονομία με επιχειρηματικό τρόπο και με καινοτομία. Μπορείτε αυτό να μου το σχολιάσετε. Βλέπετε ότι αυτό θα ήταν μια μεγάλη πηγή για την αντιμετώπιση κάποιων από αυτές τις αλλαγές. Γιατί η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μόνο από τον κρατικό τομέα, αλλά και από το πλευρά ε, των ε, επιχειρήσεων. Έπειτα, συλλογικές διαπραγματεύσεις που είπατε και κοινωνικός διάλογος. Έχουμε συστάσεις ανά χώρα στον τομέα και ενισχύουμε το κοινωνικό διάλογο και, ναι, και εσείς ε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, παρακολουθείτε το τι γίνεται με τη βάση των συμβάσεων. Οπότε, πώ θα μπορούσατε κι εσεί να μα απαντήσετε. Υπάρχουν όμω δυσκολίε στι συλλογικέ διαπραγματεύσει και ορισμένοι επιχειρηματίε φοβούνται. Και αυτό που συμβαίνει από καιρού ει είναι ότι τα κράτη-μέλη στην ουσία πέφτουν στην παγίδα όπου το κράτος ανταλλάσσει απόψεις με το εκπροσώπους των εργαζομένων και ε, με τους εκπρόσωπους των εργοδοτών. Υπάρχουν ε, κράτη-μέλη που λειτουργούν έτσι και άλλα όπου αυτό δεν υπάρχει πια. Πώς μπορούμε λοιπόν να αφαιρέσουμε την, την ιδεολογία αυτή. Γιατί οι συλλογικέ διαπραγματεύσει σχετίζονται με συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ιδεολογία, ενώ απορρίπτονται από εκείνου που υποστηρίζουν άλλε ιδεολογίε. Έχετε μια υπόψη σα κάποια πιο ουδέτερη ε, ιδεολογικά διαπραγμάτευση, μήπως δηλαδή ουδέτερα θα μπορούσαμε ε, να ξεπεράσουμε τέτοιους υφάλους ε, πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Πρώτα ο κύριος Σκαρπέτα και μετά ο κύριος Κόλλερο. Σα Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Πρώτον, για την οικονομία, μάλιστα. Βεβαίως, όπως είπα και προηγούμενα, ο πληθυσμός του ευρωπαϊκού ε, γυράσκει. Γιατί το ποσοστά θνησιμότητας μειώνονται, αλλά και ταυτόχρονα ζούμε περισσότερα χρόνια και με καλή υγεία κατά μέσο όρο. Ορισμένοι μπορεί να μην φτάνουν στα γερατιά, σε καλή και έπειτα τα τελευταία ε, χρόνια ζωής είναι συνήθως εντατικής ε, ε, φροντίδας. Ο τομέας λοιπόν της ε, φροντίδας είναι αυτός ο οποίος αναπτύσσεται και θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Μέχρι στιγμής στις περισσότερες χώρες ε, αυτή την φροντίδα την αναλαμβάνουν οι οικογένειες. Συχνά οι γυναίκες μένουν στο σπίτι χωρίς αμοιβή και φροντίζουν για τους ηλικιωμένους της οικογένειας όπως και για τα παιδιά. Ε, θα πρέπει αυτή η ευθύνη να μεταφερθεί σε ένα σύστημα όπου οι αμοιβέ θα είναι επαρκείς για τους εργαζόμενους και ταυτόχρονα θα είναι ένας τομέας που μπορεί να εκμεταλλευτεί όλο το δυναμικό και τη ζήτηση που υπάρχει. Μέσω λοιπόν ρυθμίσεων, μέσω ε, κατάρτισης και ε, νέας κατάρτισης να μπορέσουμε να, να προσελκύσει τους εργαζόμενους και μάλιστα σε θέσεις καλύτερης ποιότητας. Θέλουμε πόρους, κανονισμούς αλλά και προσπάθεια από πλευράς ε, των κοινωνικών εταίρων για να κατανοήσουν ποιες είναι οι προκλήσεις και αυτές οι εργασίες που δεν είναι καλές σε θέσεις αυτή τη στιγμή, πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας και κακές αμοιβέ να βελτιωθούν. Υπάρχει το δυναμικό.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 ε, μελέτες αυτές για τις ειδικέ συνθήκες εργασίας. Ε, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνη και για την κατάρτιση αλλά και για τα ωφέλη, τα κέρδη αυτής ε, της κατάστασης. Υπάρχουν διαφορές όπως σας είπα ανάμεσα στις χώρες αλλά ε, θα πρέπει να υπάρξουν και ανταλλαγέ καλύτερων πρακτικών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν. Εάν είσαι ανεξάρτητος επαγγελματίας, ο νόμος ε, περί ανταγωνιστικότητας σε προστατεύει απέναντι στους συναδέλφους του, σου απέναντι στους πελάτες. Δηλαδή δεν θα πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία περί ανταγωνισμού που είναι εξαιρετικά περίπλοκη, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται αυτή η νομοθεσία, ώστε οι ανεξάρτητοι επαγγελματίε να μπορούν να συμμετέχουν και αυτές τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Εγώ δεν μπορώ να προσθέσω και πολλά γιατί είμαστε σύμφωνοι ανάμεσα στους δύο οργανισμούς. Αλλά για τον κλάδο της φροντίδας είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης που έχει εντοπιστεί για το μέλλον. Όμως το ζήτημα προχωρά λίγο πιο βαθιά. Εμείς ως κοινωνία μπορούμε οικονομικά να στηρίξουμε ε, αυτούς τους ανθρώπους που θα φροντίζουν ε, τους ηλικιωμένους ε, και τα παιδιά να το κάνουν αυτό δωρεάν ή χρειάζεται αλλαγή της κατάστασης, να προσπαθήσουμε δηλαδή να ανταμείψουμε αυτού του είδους τις υπηρεσίες που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι υπηρεσίες χρήσιμες για την κοινωνία. Δηλαδή με μισθό, με σύνταξη κτλ. κτλ. Όπως σας είπα, το θέμα είναι πολύ βαθύ. Επίσης, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πρακτικά παραδείγματα. Ήμουνα σε ένα πάνελ στο Βερολίνο και είπε μια νεαρή κοπέλα ότι πρώτα απ' όλα έχει βαρεθεί ότι η οικονομία αυτού του ε, η κλασική βασική οικονομία δεν φέρνει ε, ε, ε, ωφέλη. Γιατί αυτά που δεν υπήρχαν στο business plan της ήταν ότι πολλοί από τους φροντιστές ήταν ε, ήδη ηλικιωμένοι άνθρωποι που ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους περισσότερο ηλικιωμένους που δεν θέλαν να ζήσουν χωρίς φροντίδα. Αυτό λοιπόν είναι μια θετική πτυχή της νέας οικονομίας. Για τις συλλογικέ διαπραγματεύσει τώρα, συμφωνώ με τον Στέφανο ότι αυτές γίνονται σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις κάθε φορά, ότι είναι θέμα επικουρικότητας και, και ούτω καθεξής. Πώς ξεφεύγουμε όμως από αυτού του είδους την ε, ε, ιδεολογία θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να, ε, εκτός από την μελέτη αντικτύπου, να σκεφτούμε το εξής, ότι αν λειτουργεί ε, ε, αλλά μια, μια συλλογική διαπραγμάτευση μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο ε, αλλά τελικά να είναι αίσιο το πέρας. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι και εργοδότες να καθίσουν και να τα βρουν χωρίς τις κυβερνήσεις. Μια από τις δικές μου εμπειρίες ήταν ότι όσες φορές έχω εγώ παίξει το διασωμεσολαβητή, είναι ότι οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες τα βρίσκουν συχνά καλύτερα χωρίς τον τρίτο εταίρο, δηλαδή την εκάστοτε κυβερνήσει στι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Επίσης θα πρέπει οι, οι, οι οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Πολύ ενθαρρυντικό βρήκα το παράδειγμα της Δανία, όπου μπορεί κανεί μέσω μια ψηφιακή πλατφόρμα πλατφόρμας να πάρει ε, υπηρεσίες καθαρισμού. Έχουν φτάσει σε συμφωνία συλλογική για τις μήνυμου μισθούς, τις μήνυμου ώρες εργασίας και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Ε, δεν υπάρχει και ιδεολογία. Λέμε, χρειάζεται αυτό το πράγμα και υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές. Ε, τώρα, κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας οργανώσαμε μία συνεδρίαση μαζί με την ETUC, το Διεθνή Ομοσπονδία Συνδικάτων, και εκεί ε, μίλησαν για μία οδηγία περί συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ενδιαφέρουσα ιδέα. Ξέρω ωστόσο ότι μπαίνει εκεί η επικουρικότητα, ότι είναι δύσκολο το θέμα, αλλά ίσως και εκεί θα έπρεπε να κινηθούμε προς τα εκεί με στόχο να έχουμε στην ουσία κάτι που να βγάζει νόημα και να ξανα φτιάξουμε την εικόνα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Και η επόμενη ερώτηση είναι της κυρίας Ραφάσκα που είναι η συντονίστρια του ECR. Ε, wszystko to, co dzieje się na rynku pracy jest niezwykle ciekawe i pasjonujące i nie możemy... Ο κόσμος της εργασίας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ε, και συναρπαστικός. Ε, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για εξέλιξη της αγοράς, αλλά για επανάσταση, η ρομποτοποίηση, η αυτοματοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά τα στοιχεία αλλάζουν ε, εκβάθρον την αγορά εργασίας. Και Μπορεί κανείς ε, να έχει την εντύπωση πως ορισμένοι εργαζόμενοι ε, αισθάνονται αποκλεισμένοι από αυτά τα φαινόμενα γιατί δεν καταφέρουν να συμβαδίσουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και οι ίδιοι αυτό το θεωρούν ε, μέγα κίνδυνο, την εξέλιξη δηλαδή της τεχνολογίας. Επιπλέον ε, βλέπουμε πως υπάρχουν μεγάλες ε, αποκλίσεις ε, εδαφικές. Ωστόσο, η αυτοματοποίηση ή εσείς πιστεύετε ότι δημιουργεί περισσότερες θέσεις απασχόλησης ή καταστρέφει θέσεις απασχόλησης. Πρώτη ερώτηση. Έπειτα, σήμερα αναφέρθηκε η Γαλλία και οι λύσεις οι οποίες είναι ευνοϊκές για τους εργαζόμενους. Εγώ θέλω να αναφέρω το παράδειγμα της Πολωνίας και των ατυπικών μορφών εργασίας. Υιοθετήθηκαν εθνικά μέτρα για την υπεράσπιση των εργαζομένων. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά το 2017 ε, εισήχθη το minimum ε, ορομίσθιο. Και έπειτα, για τους ανθρώπους οι οποίοι προσλαμβάνονται με άτυπα ε, συμβόλαια, άτυπες συμβάσεις εργασίας, να μπορούν να προσχωρήσουν στα συνδικάτα. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε και τον αριθμό των ανεξάρτητων επαγγελματιών και τον αριθμό των ατυπικών συμβάσεων. Και έπειτα αναφέρθηκε και η περίοδος η μεταβατική. Μα πόσο διαρκεί αυτή η μεταβατική περίοδο. Εγώ έχω την εντύπωση πως αυτή η περίοδος παρατείνεται επάπειρον, επαόριστον. Προς χάρην ευελιξίας. Και έτσι χάνεται η αίσθηση της βεβαιότητας, της ασφάλειας. Κυρίως όσον αφορά τους ε, παλαιότερους, τους αρχαιότερους εργαζόμενους. Εργαζόμενους που γνωρίζουν σήμερα πως θα πρέπει να μαθαίνουν ολόκληρη τη ζωή τους, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης που έχουν. First, Mr. Scarpetta, and then Mr. ο κύριος Σκαρπέτα και μετά ο κύριος Κόλλερ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σα την ερώτηση. Το πρώτο κομμάτι δεν το άκουσα πολύ καλά, αλλά αν σας κατάλαβα καλά να προσπαθήσω να απαντήσω. Κοιτάξτε, για να κάνουμε εικασίες ε, για το μέλλον. Αν δούμε το τι συμβαίνει τα τελευταία 10-15 χρόνια, βλέπουμε πως ε, ο ψηφιακό μετασχηματισμός και η άλλη τάση που ανέφερα πριν αλλάζουν ε, με κέριο τρόπο την αγορά εργασίας. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και χώρες του ΩΣΑ βλέπουμε τη λεγόμενη πόλωση της αγοράς εργασίας, δηλαδή πολλές δουλειές δημιουργούνται στο υψηλό επίπεδο και απαιτούν πολλές δεξιότητες, αλλά και πολλές στο χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων ε, και σταδιοδρομίας. Και στη μέση, όπου ήταν οι περισσότερες δουλειές στο παρελθόν, έχουμε ε, μείωση των θέσεων εργασίας. Οπότε δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας, αλλά δεν είναι όλες της ίδιας ποιότητας. Κάποιες έχουν χαμηλό επίπεδο μάλιστα, λόγω των συμβάσεων, λόγω της πληρωμής ε, και λόγω ε, των προοπτικών σταδιοδρομίας. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που κινδυνεύουν ε, να διολυστήσουν σε μια, ποιότητα, σε μια δουλειά χαμηλής ποιότητας να μετακινηθούν προς τα πάνω. Υπάρχει γεωγραφική διάσταση εντός των χωρών και μεταξύ των χωρών, αλλά και κλαδική διάσταση και ηλικιακή διάσταση, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για τους νέους να μετακινηθούν προς τα επάνω, καμιά φορά πιο δύσκολο για έναν μεσήλικα. Ναι, οπωσδήποτε. Η Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές και μη χώρες έχουν εφαρμόσει διάφορες μεταρρυθμίσεις και προτείνω να δείτε την έκθεση που δημοσιεύσαμε πριν από κάτι μήνες που βασικά είναι μια συλλογή των απαντήσεων που δώσαν οι χώρες σας ε, όσον αφορά τις απαντήσεις στις νέες μορφές εργασίας και είναι εκπληκτικό το πώς έχουν κάνει οι χώρες ήδη για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ε, που συζητάμε σήμερα στον ΩΣΑ. Κάποιες από αυτές τις απαντήσεις αφορούν βεβαίως συγκεκριμένα τις ανάγκες αυτές, αλλά υπάρχει και κάποια συνοχή στα μέτρα αυτά. Προσπαθούμε να κλείσουμε αυτό το κενό, πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, ε, κατάρτιση και επανακατάρτιση. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω όταν μιλάμε για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες ε, οι εξαρτώμενους, αν θέλετε, ελεύθερους επαγγελματίες, οι χώρες αντιρούν διαφορετικά και οι εταιρείε ε, των πλατφορμών είναι πολυεθνικές και το ότι δεν υπάρχει ακριβώς ε, ενιαία αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή τόπου εγκατάστασης. Θεωρώ ότι εντό Ευρώπη θα πρέπει να γίνει ένας διάλογος για το πώς θα ρυθμιστεί ε, η αγορά αυτή η οποία αυξάνεται. Στο δεύτερο θέμα είναι οι άτυπες ε, μορφές ε, εργασίας. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι έκανε κάποιες μεταρρυθμίσεις η Πολωνία και εδώ πέρα ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μπορούν να πάνε όλοι σε τις τυπικές συμβάσεις αορίστου διαρκείας. Το θέμα είναι ποια θα είναι η απάντηση της νομοθεσίας της ρύθμισης για να διατηρηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας και να μην αποτελέσουν ένα βήμα, θέλετε, σε καλύτερες ε, θέσεις. Είναι θέμα λοιπόν φορολογίας, συνθήκων εργασίας. Πολλά λοιπόν πρέπει να γίνουν για τις ε, μη τυπικές μορφές εργασίας για να γίνουν καλύτερες. Και εδώ πέρα λοιπόν έχουμε έναν κλάδο που μπορεί να αναλυθεί δράση. Τέλος. Σε κάποιες χώρες έχει υπάρξει σημαντική αύξηση στην αυτοαπασχόληση γιατί υπάρχουν ισχυρά κίνητρα επίσης για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να είναι αυτοαπασχολούμενοι γιατί υπάρχει ουσιαστική διαφορά ε, στη φορολογία. Μπορούμε να μειώσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ των διαφόρων μορφών απασχόλησης. Ευχαριστώ. Και πάλι για να συμπληρώσω τις ε, παρατηρήσεις αυτές αυτό το οποίο είπατε για την ε, μεταβατική περίοδο η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Ναι, ναι, πράγματι αυτό συμβαίνει. Το πρόβλημα είναι ήδη από το σχολείο. Πώς προετοιμάζουμε τους ανθρώπους ε, για μια διαρκή μετάβαση. Πώς θα έχουν την αίσθηση ότι δεν θα είναι εγκαταλελειμμένοι και αφήγει φύγει αυτό, αυτή η αίσθηση της ανασφάλειας. Και εκεί από την σκοπιά του ΑΕΛΟ θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο στήριξης. Όχι μόνο οι ε, κρατικές υπηρεσίες εργασίας, αλλά ε, κοινωνική προστασία στην περίπτωση στην οποία πρέπει να υπάρξει μετάβαση από τη μία δουλειά στην επόμενη. Μια καλή ανάλυση της αγοράς εργασίας ε, και το που θα χρειάζονται βεβαίως ε, μελλοντικά οι δεξιότητες σου. Γιατί είναι πολύ απογοητευτικό το να εκπαιδεύεσαι και να μην σε χρειάζεται αγορά εργασία. Λοιπόν, πολλές χώρες ε, και η Πολωνία, το αναγνωρίζω αυτό, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Το άλλο είναι αυτό το οποίο είπατε, κοινωνικά δικαιώματα ανεξαρτήτως καθεστώτος. Αυτό αφορά ακριβώς και την ε, οικονομία αυτή των πλατφορμών ε, και οι άνθρωποι που εργάζονται με αυτή τη μορφή έχουν κάποια γενικά δικαιώματα όπως επίδομα ανεργίας, ασφάλιση υγείας, σύνταξη, αλλιώς ε, δεν θα χάσουν ποτέ αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας και αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων των μελών της Επιτροπής μας πρώτα θα κάνετε τις ερωτήσεις και μετά θα δώσουμε τον λόγο στους προσκεκλημένους μας. Η κυρία Σπάρανταγκ λοιπόν και ο κύριος Μάντερς να ετοιμάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και για την παρουσίαση σας. Έχω μία ερώτηση γιατί ε, παρουσιάζεται μία ατζέντα μετάβασης για ένα μέλλον που θα λειτουργεί για όλους και είπατε ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες τάσεις και παραδείγματο χάρη η ρομποτοποίηση μπορεί να επηρεάζει το 17% των εργαζομένων αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρη για το πού βρίσκεται η αγορά εργασίας καθώς θεωρώ ότι εγώ θεωρώ ότι το 100% των ανθρώπων θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή και δεν ακούω τίποτα για τη μετάβαση που θα υπάρξει, την αλλαγή των θέσεων εργασίας και τη μεγάλη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία και αναρωτιέμαι γιατί δεν περιλαμβάνεται και πώς ε, δεν υπάρχουν αυστηρές ε, ε, συστάσεις πολιτικής γιατί βεβαίως κάποιοι θα πρέπει να το πληρώσουν αυτό το κόστος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντερς και η κυρία Ντούρα Φερνάντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ Εκπροσωπώ το κόμμα των ηλικιωμένων από την Ολλανδία 50 ετών και πάνω, δηλαδή μιλάμε για το μισό πληθυσμό αυτή τη στιγμή. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, στις συστάσεις σας δεν βλέπω τον υγιεινό τρόπο ζωής, γιατί αν να χρησιμοποιήσουμε την ε, γύρια οικονομία, θα πρέπει ο κόσμος να είναι υγιής και αν δεν εστιάσουμε σε αυτό τελικά η ασφάλιση υγείας θα γίνει πάρα πολύ ακριβή και δεν μπορούμε να ζητάμε από τον κόσμο να δουλεύει μέχρι να είναι 70. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει φτάσει η στιγμή να ξανασκεφτούμε γιατί τώρα ζητούμε λύσεις ε, με παραδοσιακό τρόπο και τα λοιπά, τα συνδικάτα και τα σχετικά. Αν δω τον αριθμό σας που υποθέτω ότι είναι του 2016, είναι ήδη 2-3 ετών, η ζήτηση για τα ρομπότ αυξάνεται κατακόρυφα και ποτέ κανείς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ένα ρομπότ ως ε, άνθρωπος ε, στην παραγωγικότητα. Έχει φτάσει η στιγμή να ξανασκεφτούμε νέους τρόπους διακυβέρνησης γιατί κομμουνισμός, ε, σοσιαλισμός, καπιταλισμός, ε, τα ξέρουμε και τελικά με αυτούς τους αριθμούς ε, τίποτα από αυτά δεν θα λειτουργήσει στο μέλλον. Θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος διακυβέρνησης, αλλιώς σβήνει το μικρόφωνο του Μουλτή. Γιατί τελικά οι διοκτήτες των ρομπότ θα αποφασίζουν τα πάντα και δεν νομίζω να είναι αυτό, αυτό το οποίο θέλαμε. Ίσως την επόμενη φορά μπορούμε να προσκαλέσουμε και απευθύνομαι στην κυρία Πρόεδρο, τον κύριο Πικετή, ο οποίος έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για το μέλλον της οικονομικής σκέψης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Φερνάντες δεν θέλει να κάνει ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται, λέει η κυρία Φερνάντες, γιατί έγινε η ερώτηση που ήθελα να κάνω. Οπότε μένει η κυρία Σόιμπη. Είστε έτοιμοι. Ωραία. Και... Και να ετοιμάζει ο κύριος Κάνιεφ. Καλημέρα. Ερώτησή μου απευθύνεται στον κύριο Σκαρπέτα. Ενδιαφέρθηκα πολύ για αυτό που είπε στην εργασία σας για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες. Ελπίζω η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων, να έχει δυνατότητα να επεξεργαστεί την επόμενη οδηγία για τις πλατφόρμες όπου εκεί επανειλημμένα τίθεται το θέμα στις συνεδριάσεις μας. Αναφερθήκατε στην ανάγκη καταπολέμησης των ανεξαρτήτων να προσφέρουμε περισσότερη κοινωνική προστασία στους εργαζομένους στις πλατφόρμες και αναφερθήκατε στο ότι, όπως είπατε, θα πρέπει να φεύγουμε νέους, ε, νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου. Για τους εργαζομένους των πλατφορμών, ερώτηση. Περί τίνο πρόκειται. Θα πρέπει στου εργαζομένου των πλατφορμών να μπει ο κοινωνικό διάλογο με κλασικό μοντέλο. Έχουμε από τη μία πλευρά του εκπροσώπου των πλατφορμών και από την άλλη πλευρά του εκπροσώπου των εργαζομένων. Ή αναφέρεστε σε εφεύρεση νέων μορφών κοινωνικού διαλόγου, διότι έχετε υπόψη άλλα μοντέλα που ίσω είχαν ε, ε, αποτελέσει αντικείμενο πειραμάτων κάπου. Εν τη αυτή περιπτώση θα ήθελα να γνωρίζω περισσότερα αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Εγώ όταν θέλω να παρακινήσω το γιο μου να διαβάσει μαθηματικά, του λέω ότι όταν θα μεγαλώσει θα υπάρχουν δύο ειδών δουλειές. Ε, είτε θα προγραμματίζει ρομπότ, είτε θα καθαρίζει ρομπότ. Οπότε αν δεν θέλει να καθαρίζει τα ρομπότ πρέπει να μάθει να τα προγραμματίζει. Αλλά σοβαρά τώρα νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στην διάγνωση. Αλλά αυτό το οποίο ακούω εγώ από σας ως αντιμετώπιση είναι ε, η αύξηση είναι πράγματα τα οποία αυξάνουν το κόστος ε, εργασίας ε, δουλειών που είναι ήδη πολύ ακριβές και για τους εργαζόμενους και για τους αυτοαπασχολούμενους. Δεν είναι πιο σωστό ειδικά εν ώψη της πράσινης μετάβασης να βρεθεί ένας τρόπος να μειωθεί δραστικά το κόστος ε, για τους εργαζόμενους εκείνους που χρειάζονται νέες δεξιότητες ε, για να γίνει η μετάβαση, για όσους χρειαστεί να κάνουν αυτή τη ε, μετάβαση. Για το 90% εργαζομένων και εργοδοτών. Σας ευχαριστώ θα ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο απαντήσεων με τον κύριο Κόλερ. πρώτη ερώτηση. Δεν μιλήσαμε για τη δίκη μετάβαση σε πράσινες ε, θέσεις εργασίας στην παρουσίασή μου. Είπα ότι η δίκη μετάβαση σε πράσινες δουλειές ήταν στο μίσο που στο μέλλον ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τις εργασίες και θα πρέπει να βοηθήσουμε τη μετάβαση να δώσουμε δυνατότητα αναβάθμιση δεξιοτήτων σε εκείνου που πάνε σε πράσινε δουλειέ. Και υπάρχουν πολλές δυνατότητες να έχουμε κέρδη, αύξηση θέσεων εργασία μέσω των πρασίνων θέσεων εργασία. Είμαστε, το ξέρουμε αυτό, για την υγιεινή, τον υγιεινό τρόπο ζωής. Ποιο είναι το πρόβλημα όσον αφορά το ILO. Το βλέπουμε από την άλλη πλευρά. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος δεν αρρωσταίνει όταν εργάζεται. Οπότε η υγιεινή και ασφάλεια στην απασχόληση. Πρώτα, οι φορείς υγείας εξετάζουν τις πτυχές υγείας. Όμως η ατζέντα για το 2030 είναι ένας τρόπος να ξεπεράσουμε αυτή την απομονωμένη ανάλυση των θεμάτων. Συνεργαζόμαστε στενά λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εξετάσουμε και τις δύο όψεις και ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πιστεύω. Τούτου λεχθέντος, ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι η αύξηση της διάρκεια ζωής και ενεργάζονται μέχρι πιο μεγάλη ηλικία κάποιοι. Εάν αυξήσουμε λοιπόν το όριο συνταξιοδότησης, τότε πρέπει να εξασφαλίσεις ότι η δουλειά ή ο τόπο εργασία ταιριάζει για πιο ηλικιωμένους ανθρώπου για να εργάζονται επί μακρότερων. Αυτό εξετάζουμε. Και έχουμε κάνει κάποιες σχετικές προτάσεις. Κυβερνήσεις και ρομπότ. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι, μας κυβερνούν τα ρομπότ ή εμείς κυβερνάμε τα ρομπότ. Εγώ νομίζω ότι το δεύτερο μάλλον ισχύει. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ρομπότ σε τομείς που μας είναι χρήσιμο. αλλά εργάζεται και με το κόστος εργασίας. Το κόστος εργασίας είναι πολύ ψηλό για χειρονακτική εργασία που πρέπει να έχουμε ρομπότ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μας ελέγχουν τα ρομπότ. Πρέπει να βρούμε άλλες μορφές εργασίας. Όχι μόνο για, να, για καθαρισμό ρομπότ κλπ. Παράδειγμα. Μ' αρέσουν τα παραδείγματα. Πήγα στο πρωτάθλημα δεξιοτήτων, ανθρωπίνων δεξιοτήτων στο Καζάν, στη Ρωσία. Είχαν 60 επαγγέλματα. Θέμα. Κλασική εργασία, πώς να τη συνδυάσει με τα ρομπότ. Εντυπωσιάστηκα. Βλέπω ότι είσαστε καλοντιμένοι. Εντυπωσιάστηκα από ένα ράφτη που με έσπρωξε σε μία μηχανή σάρωσης, μου πήρε τα μέτρα το ατελές μου σώμα μετρήθηκε, ούτω ώστε αν θέλω να παραγγείλω κάτι μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, τότε έχω μία app, μία εφαρμογή και έχουν τα μέτρα μου και έχω τα ρούχα μου. Η αντίληψη των ρομπότ είναι πολύ στενή. Πρέπει να διευρύνουμε την αντίληψή μας περί ρομπότ. Και όσον αφορά τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση αυτών. Υπάρχουν ενδιαφέρουσε ιδέε που δεν έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Γίνεται συζήτηση, Φερρυπίν, σε κάποιε χώρε. Τι συζητάνε. Ένα ρομπότ αντικαθιστά ένα εργαζόμενο. Πρέπει να φορολογηθεί το ρομπότ όπω φορολογεί ένα εργαζόμενο. Ενδιαφέρουσα έννοια αυτή. Το άλλο ερώτημα τώρα. Αύξηση του κόστους εργασίας εκπαίδευση, κατάσταση, αναβάθμιση δεν πρέπει να θεωρείται κόστος, πρέπει να θεωρείται επένδυση. Πρέπει αυτή την επένδυση να τη λαμβάνει υπόψη και να μπαίνει και στον προπολογισμό σαν επένδυση και όχι κόστος. Οπότε αύξηση του κόστους εργασίας στο θέμα αυτό κάπως αλλάζει. Ευχαριστώ πολύ. Έξοχες ερωτήσεις, λέει και ο Σκαρπέτα. Πολύ γρήγορα. Πολλά υπόθηκαν για τη δίκαιη μετάβαση. Είναι μία από τις βασικές μεγάλες τάσεις. Δεν αναφέρθηκα στο τι αντίκτυπο έχει στην αγορά εργασία, αλλά ότι θα παραγάγει νέε θέσει απασχόληση. Η φύση τη εργασία εξαρτάται τι είδου μετάβαση θα γίνει, καθαρή ενέργεια κλπ. Τα βασικά χαρακτηριστικά όμως της δουλειάς, στις νέες δουλειάς δεν θα διαφέρει τόσο με τεχνολογία, θα, θα αλλάξουν κάποιες δεξιότητες ο τόπο εκτέ εργασία, αλλά θα επηρεαστούν όλα αυτά από τη γύρανση και την ψηφιακή μεταμόρφωση και από την ολοκλήρωση και ενοποίηση των οικονομιών μα. Είναι μία από τι μεγάλε τάσει που θα διαμορφώσει μέσω μακροπρόθεσμα δραματικά το μέλλον μα, αλλά όσον αφορά την αγορά εργασία. Πράσινε θέσει εργασία διαφέρουν πολύ από τι παλιέ. Το μελετήσαμε πολύ όσον αφορά δεξιότητα και γνώσει, αλλάζει η τοποθεσία, χαρακτηριστικά κλπ. Για τον υγιεινό τρόπο ζωής. Και στον τον λέμε το θέμα της υγείας. Τι σημαίνει, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα και κοινωνίε στη διάρκεια του βίου εργασία, πρέπει να δράσουμε, επενδύοντα περισσότερα σε πρόληψη από ασθένειε και πολύ πιο πριν. Κάποια θέματα υγεία που αναφέρατε ισχύουν, διότι δεν δαπανούμε πολλά στην πρόληψη έχουμε μειώσει στην πρωτοβάθμια μέρημνα τα χρήματα και εξοδεύουμε περισσότερα σε νοσοκομεία και σε άλλες μορφές φροντίδας εντός αγωγικών. Στην παγκόσμια κρίση ένας τομέας δημοσίας δαπάνης υγείας ε, ε, επηρεάστηκε κατά πολύ η πρόληψη. Οι άλλοι τομεί έκαναν μικροπροσαρμογές αλλά η... χτυπήθηκε ιδιαίτερα η πρόληψη και τι δεξιότητε. Αν θέλουμε να αποφύγουμε τα άτομα να μην μπορούν να προσαρμοστούν στι δεξιότητε, πρέπει να επενδύσουμε μάλλον για να προσαρμοστούν σε όλη τη, στη διάρκεια του κύκλου παιδείας να τους ε, να παρεύουμε και να δώσουν δυνατότητα διαβίου εκπαίδευση. Για την υγεία και τη γύρανση. Εγώ αναφέρθηκα και στο προσδόκιμα ζωή. Ζούμε περισσότερο, αλλά δεν ζουν όλοι με καλή υγεία σε μεγάλη ηλικία. Και γι' αυτό χρειάζεται και η πρόνοια και επένδυση για πρόληψη και υποστήριξη να ληφθούν υπόψη. Για τα ρομπότ που παίρνουν τη δουλειά μα, τι δουλειέ μα. Σα είπα ποια είναι η αξιολόγησή μα. Ποιο είναι το βασικό θέμα και μπορούμε να κάνουμε πολλά. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Στον ΩΣΑ μας δόθηκε εντολή, έχουμε παρατηρητήριο για τη τεχνητή νοημοσύνη. Να αναλύσουμε περί τίνος πρόκειται. Η τεχνητή νοημοσύνη που βρίσκεται σήμερα. Τι δυνατότητες υπάρχουν να προχωρήσουμε. Τεχνολογικά τι δυνατότητες υπάρχουν. Διοντολογικά τι γίνεται για τη χρήση αλγορίθμων και εκμάθηση από μηχανέ τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα στι προσλήψει χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιούν την αξιολόγηση τη επιδόση των εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη και στο μέλλον θα γίνεται αξιολόγηση ε, οι δυνατότητε των ατόμων, οι ανάγκε του κλπ. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, τι δυνατότητε προσφέρει και πώ παρεμβαίνει η νομοθεσία για να πλαισιώσει το θέμα. Για του εργαζόμενου σε πλατφόρμες, καλή ερώτηση συλλογικέ συμβάσει, αν θα χρησιμοποιήσουμε παραδοσιακέ συλλογικέ διαπραγματεύσει ή όχι. Εργαζόμενοι σε πλατφόρμε είναι διαφορετικοί εργαζόμενοι. Οδηγό ταξί. Έχει συναλλαγή μεταξύ πελάτη και αυτού. Και, μέσω παραδο... και πλατφόρμα, αν γίνει, παραδοσιακή δουλειά. Άλλο, άλλη μορφή εργασία είναι οι ψηφιακέ υπηρεσίε που παρέχουν ψηφιακά εργαλεία σε κάποιον που θέλει να τα χρησιμοποιήσει όχι όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες θέλουν να θεωρηθούν εργαζόμενοι, θέλουν να θεωρηθεί ότι έχουν ένα βαθμό αυτονομίας. Αλλά επαναλαμβάνω σε πολλές χώρες, αν είσαι ανεκράτος εργαζόμενος, δεν μπορείς να πραγματευτεί με τους ομοτήμους σου και με τους πελάτες σου και με αυτούς που αγοράζουν τις υπηρεσίε σου. Να επιτρέψουμε σε εργαζόμενο σε πλατφόρμα να, να διαπραγματευτεί συνθήκες εργασίας και αμοιβέ είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να προσφέρουμε όλα τα πακέτα όπω ένα μισθωτό φερειπίν σε κάποιε χώρε επεκτείνεται η κοινωνική προστασία και ελάχιστο επίπεδο κοινωνική προστασία στου εργαζόμενου σε πλατφόρμε και σε πολλέ ε, ευρωπαϊκέ χώρε. Η αύξηση του κόστου εργασία. Ενδεχομένω, δεν ξέρω όμω. Ε, κατάρτιση, Φερρυπίν. Κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε δαπανούν πολλά χρήματα για την κατάρτιση. Πολλά χρήματα. Στη Γαλλία 55 δισεκατομμύρια για τεχνική ε, επαγγελματική κατάρτιση αυτά τα χρήματα πώς χρησιμοποιούνται και ποιος έχει πρόσβαση στους πόρους. Αυτό είναι το θέμα. Η Γαλλία πάει σε λογαριασμό εξατομικευμένων. Έχουν το δικαίωμα για κάποια χρήματα που θα χρησιμοποιήσει για κατάτηση. Η μεγάλη πρόκληση εδώ και σε άλλε χώρε όπω η Ολλανδία είναι να εξασφαλίσουν ότι αυτοί που έχουν τα χαμηλέ δεξιότητε να έχουν κατάλληλα εργαλεία να το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά. Η κοινωνική προστασία να καλύπτει πράγματι μπορεί να κοστίζει περισσότερα χρήματα. Αλλά αν σκεφτούμε κάποιου από του εργαζόμενου σε πλατφόρμε, εφόσον είναι εξάρτητοι εργαζόμενοι, δεν πληρώνουν τις ίδιες κοινωνικές εισφορές. Σε κάποιες, περιπτώσεις, σε υπάλληλο, οπότε ε, ζητούν από την εταιρεία να πληρώσει μια ελάχιστη κοινωνική εισφορά, ε, κοινωνικής ασφάλισης μάλλον. Εγώ αναφερόμουν στο θεματολόγιο, στην ατζέντα τη μετάβαση. Κάποιοι πόροι μπορεί να προσθέτουν απάσει πρωτοβουλίε που σχετίζονται με τη διαχείριση τη ψηφιακή μετάβαση. Τα BEPS, ε Φερρυπίν αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τη φορολόγηση είναι γενικές πρωτοβουλίες που μπορούν δημιουργήσουν ένα εισόδημα που ίσως να φορολογηθεί σωστά, που παράγει εισόδημα και να βοηθήσει αυτούς που δεν έχουν αρκετούς πόρους για να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή, αυτή τη μετάβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να κλείσω το πρώτο τμήμα του σεμιναρίου μας, να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ και μας κάνατε τόσο ζωντανές ε, εισηγήσεις. Οφείλω να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη με τις απαντήσεις που μας δώσατε σε όλες μας τις ερωτήσεις, διότι αναφέρατε όλες τις προτεραιότητες με τις οποίες ασχολούμαστε στο χαρτοφυλάκιο και στην Επιτολή Απασχόλησης. Είναι καλό να ακούμε ε, συζητήσεις που βασίζονται στα στοιχεία για τα θέματα τα οποία τόσο μας απασχολούν. Κάποιες φορές δεν έχουμε αρκετά στοιχεία εσείς όμως σήμερα είστε εδώ και μπορείτε να μας δώσετε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στις προκλήσεις που μας περιμένουν όσον αφορά τη μακροχρόνια φροντίδα, τη δραστήρια γύρανση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις κοινωνικά αποκλεισμένες κοινότητες για το πόσο πόσες δεξιότητες έχουν οι άνθρωποι που περιμένουμε να επιτύχουν στις ανοιχτές αγορές εργασίες και όλα όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Dear colleagues, uh, let me open the second part. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ε, περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος ε, του εργαστηρίου, ε, το θέμα το οποίο μας απασχολούσε, η, διεθν, η εγγύηση για τα παιδιά. Όλο την συζητάμε, αλλά δεν ξέρουμε τι μορφή έχει και τι μορφή θα πρέπει να έχει. Οπότε, Ας ε, καλωσορίσω την κυρία Μέρι Ντέιλι. του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης ε, που θα μας μιλήσει για το θέμα της καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας. Καλώς ορίζουμε λοιπόν την κυρία Μέρι Ντέιλι Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα να μιλήσω για την ε, εγγύηση για τα παιδιά και να ευχαριστήσω το αρμόδιο τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντός 15 λεπτών ελπίζω να είμαι αρκετά σύντομη και ο βασικός μου στόχος είναι να εκθέσω αυτό το οποίο θεωρώ εγώ ως ιδιαιτερότητες ε, της εγγύησης για τα παιδιά, ειδικά σε σχέση με την σύσταση για να επενδύσουμε στα παιδιά. Και στο τέλος της παρουσίασής μου θα κάνω κάποιες προτάσεις για το πώς θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε την εγγύηση αυτή. Και να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το φόρουμ και οπωσδήποτε η εγγύηση αυτή ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως ε, το φόρουμ και το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα να συμπενθυμίσω ότι έχουμε πρόβλημα παιδικής φτώχειας ε, στην Ένωση. Ένα 25% των παιδιών, 24 εκατομμύρια παιδιά στην Ένωση δηλαδή ζουν ε, στον ορισμό της φτώχειας, δηλαδή είτε κάτω από μια γραμμή φτώχειας ή σε νοικοκυριά με ουσιαστικές ηλικές ε, ελλείψεις ή με χαμηλή ένταση εργασίας. Νομίζω όλοι συμφωνείτε ότι είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός για μια τόσο πλούσια περιοχή του κόσμου. Ναι, είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα. Γνωρίζουμε ποιε είναι οι χώρες που έχουν του υψηλότερου αριθμούς παιδικής φτώχεια, αλλά σε κανένα κράτος μέλος δεν είναι λιγότερο από 14-15% οπότε εγώ θα έλεγα ότι είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα που πρέπει να δει κάθε χώρα και θα δείτε στην διαφάνεια της χώρες με το υψηλότερο και το χαμηλότερο ποσοστό. Βεβαίως ε, τα ποσοστά μειώνονται και αυτό είναι θετικό, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για την ερμηνεία, γιατί πραγματικά συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της ανάκαμψης ε, με, από την μεγάλη ύφεση. Θα ήθελα τώρα να πω λίγα λόγια για το πώς θα πρέπει να ερμηνεύσουμε την παιδική φτώχεια. Νομίζω ότι υπάρχει μια ε, συμφωνία μεταξύ πολιτικών και πανεπιστημιακών ότι είναι ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα και η εγγύηση για τα παιδιά το αναγνωρίζει αυτό με τους πέντε γίγαντες όπως τους λέω εγώ δηλαδή επαρκής διατροφή, αξιοπρεπής στέγαση, ε, δωρεάν παροχή υγείας, ε, εκπαίδευσης και προσχολικής εκπαίδευσης. Οπότε ήδη υπάρχει κάποια αναγνώριση των βασικών στοιχείων ε, της ε, πολυεπίπεδης ε, διάστασης της στόχιας παιδιών και ενηλίκων. Γνωρίζουμε ότι η φτώχεια στην παιδική ηλικία επηρεάζει ολόκληρη τη ζωή τους και τις συνθήκες στις οποίες ζουν και το μέλλον τους. Και είναι μια πηγή ανισότητα και στο παρόν αλλά και στο μέλλον μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για τους ε, κινδύνους, ε, τους παράγοντες κινδύνου, ε, τη φτώχεια και ειδικά την παιδική φτώχεια. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι το επίπεδο εκπαίδευση των γονιών ο οποίο ξεπερνάει όλους τους άλλους παράγοντες όπως τον ανήκει κανείς σε μειονοτική ομάδα ή να είναι μετανάστηση το να μην εργάζονται οι γονείς. Υπάρχουν Δύο μηνύματα λοιπόν που θα ήθελα να περάσω εδώ πέρα. Το ένα είναι ότι απαιτούνται διάφορες πολιτικές και το δεύτερο είναι ότι είναι κάτι το οποίο έχει και θετικές πτυχές γιατί γνωρίζουμε ότι με παρεμβάσεις μπορούμε να μειώσουμε την παιδική φτώχεια εδώ και τώρα και τις μελλοντικές συνέπειες. Τώρα θα αναφερθώ στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το ότι οφείλουμε να πούμε ότι η παιδική φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός ε, είναι θέμα κυρίως των κρατών μελών και πρέπει να το πούμε αυτό. Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών γενικώ. Όμως αυτό βεβαίως δεν σταμάτησε την Ένωση από το να παίξει ηγετικό ρόλο και Υπάρχουν σημαντικά επιτεύγματα, σημαντικές νέες ιδέες, μεταξύ των οποίων και η εγγύηση για τα παιδιά, τα προγράμματα και ε, νομική, τα νομικά μέσα, παραδείγματο χάρη είναι η Σύμβαση του για τα δικαιώματα του παιδιού, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και τα λοιπά. Και βεβαίως το τέταρτο βασικό στοιχείο νομίζω της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η συστάση του 2013, επένδυση στα παιδιά, να σπάσει ο κύκλος της μειονεξίας, η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδιαίτερο στο άρθρο 24, το οποίο εγγυάται τέτοιες ε, προστασίες στα παιδιά που θα τους δώσει την δυνατότητα να ε, ευημερήσεων και ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας του 2017 Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ειδικά η αρχή παριθμών 11, η οποία πέρα από το ότι εγγυάται ποιοτική και προσιτή οικονομικά ε, προσχολική φροντίδα, ε, λέει ότι τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την φτώχεια και τα πιο στερημένα παιδιά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ειδικούς πόρους για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Οπότε υπάρχει ήδη σημαντική δουλειά που γίνεται και κάτι το οποίο καθίσταται σαφές είναι οι ανάγκες ε, στόχευσης των εν λόγω παιδιών. Τώρα, στην επόμενη διαφάνεια, θα αναφερθώ σύντομα στην σύσταση του 2013 για να σας υπενθυμίσω και πάλι τι ακριβώς είναι το θέμα και το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, στην σύσταση ε, συστάθηκε στα κράτη-μέλη να εισαχθούν στρατηγικές με βάση τα δικαιώματα, ολοκληρωμένες στρατηγικές και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια ισχυρή δήλωση πολιτικής που πρότεινε ξεκάθαρες γραμμές ανάπτυξης πολιτικής και ήταν και πάρα πολύ φιλόδοξη. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Και βλέπετε εδώ στην διαφάνεια ότι υπήρχαν τρία σημεία εστιασμού επαρκής ε, πόρη και κυρίως εννοούμε για τους γονείς ε, των παιδιών και ε, αυτό πρέπει να το έχετε κατά νου. Είτε τα, παιδιά, τα μέτρα απευθύνονται προς τα παιδιά είτε προς τους γονείς είτε και προς τους ε, δύο και νομίζω εδώ είναι πολύ ιδιαίτερη η εγγύηση για τα παιδιά και είναι μια θετική εξέλιξη. Το άλλο είναι η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και το ότι οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να είναι προσβάσιμες, προσιτές οικονομικά και το τρίτο είναι πραγματικά το πετράδι του στέματος ε, των δικαιωμάτων του παιδιού, το ότι αντιμετωπίζονται ως άτομα με δικαίωμα να ακουστούν σε καταστάσεις που τους αφορούν και δικαίωμα προς την ανάπτυξή τους, ε, ειδικά σε θέματα αναψυχής κτλ. Όσον αφορά τα επιτεύγματα των συστάσεων μέχρι στιγμής, σε γενικές γραμμές ε, υπάρχουν πολλές δράσεις σε επίπεδο κρατών μελών σε σχέση με την ε, παιδική φτώχεια και πολλές δράσεις που λαμβάνονται. Πολλά παραδείγματα από τα οποία μπορούμε να διδαχτούμε. Όμως θα έλεγε κάποιος ότι ως απάντηση προς την σύσταση είχαμε μια ροή μάλλον μικρή ε, λιγότερο από ό,τι θα θέλαμε παρά το ότι είναι ακόμα νωρί. Ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε το 2013 και αν έμενε κανείς να έχει αντίκτυπο μέχρι το 2017-2018 είναι κάπως υπερβολικά φιλόδοξο. Αλλά πέρα από το επίπεδο των κρατών μελών τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν ενσωματώθηκε και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτό το βλέπουμε από την έλλειψη προσοχής που δίνεται στις ε, συστάσεις αναχώρα και στην εκταμίευση κάποιων κονδυλίων. Η εξαίρεση βεβαίως εδώ πέρα είναι το Ταμείο για την Βοήθεια στους πιο ε, ευάλωτους και εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα παιδιά υποφελούνται πάνω από 4 εκατομμύρια παιδιά το έτος είτε από τρόφιμα ε, είτε μέσω του σχολικού εξοπλισμού κτλ. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό γιατί τα παιδιά ε, στοχεύονται απευθείας εδώ πέρα. Οπότε τα αποτελέσματα είναι ότι η παιδική φτώχεια δεν λαμβάνει την απαιτούμενη προσοχή και το δίδαγμα που πρέπει να αντλήσουμε εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να το κατονομάσουμε. Αν θέλουμε να υπάρξει αλλαγή πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Να στραφώ τώρα στην εγγύηση για τα παιδιά. Τρεις ε, διαφάνειες έχω ακόμα, νομίζω ότι είμαι εντός του χρόνου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το καινούριο ως παρέμβαση σε σχέση με τις ε, συστάσεις. Οπότε βασίζεται στο ότι η σύσταση αυτή θα πρέπει να απτυχθεί και να υλοποιηθεί πλήρως. Α, ναι, ναι, έχω μείνει πόσες πίσω. Δεν, δεν προχωράει. Α, να το, να το. Λοιπόν, βασίζεται στην υπόθεση ότι η σύσταση θα εφαρμοστεί πλήρως, αλλά πηγαίνει και παραπέρα. Είναι ένα επιπρόσθετο μέσο όπως ε, το βλέπω και έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι εστιάζει στα φτωχότερα παιδιά είναι προσανατολισμένο προς αυτήν την κατηγορία παιδικού πληθυσμού και το άλλο είναι το εξής εδώ πέρα βεβαίως βλέπουμε την επιδεινούμενη κατάσταση κάποιων παιδιών γιατί αυτό το οποίο δεν συνειδητοποιούμε είναι ότι το κενό, ο βαθμός κατά τον οποίο οι άνθρωποι είναι κάτω από την γραμμή της φτώχειας ε, επιδεινώνεται για τα παιδιά και νομίζω ότι ε, βλέπει την φτώχεια ως πηγή ανισότητας. Οπότε έχει αυτές τις πέντε διατάξεις ε, και πάω αρκετά γρήγορα εδώ πέρα. Στην προτελευταία διαφάνεια βλέπετε έναν πίνακα που συγκρίνει ξεκάθαρα τις συστάσεις ε, της εγγύησης αυτής και βλέπετε ότι ενώ υπάρχουν εδώ πέρα ε, τα δικαιώματα του παιδιού, εγώ θεωρώ ότι η εγγύηση είναι κάτι το πολύ πιο στοχευμένο, π.χ. σαφώς αφορά τις υπηρεσίες, ενώ η σύσταση αφορούσε συμμετοχή και εισόδημα και απασχόληση και εστιάζει ιδιαίτερα στα φτωχά παιδιά και δίνει προτεραιότητα στα παιδιά. Οπότε εγώ θα σας έλεγα ότι υπάρχουν ε, εδώ πέρα τρεις όροι που πρέπει να πληρούνται. Πρώτον, εάν εστιάζει απευθείας στα παιδιά και όχι στους γονείς ή σε ε, θεσμικά όργανα ή σχολεία ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Δεύτερον, σε ποια παιδιά απευθύνεται και εάν εστιάζει ειδικά στα πιο στερημένα παιδιά και το τρίτο είναι εάν αφορά κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία. Είναι προσανατολισμένο σε υπηρεσίες και ειδικά την διατροφή, τη στέγαση, υγεία, εκπαίδευση ή ε, προσχολική ε, φροντίδα. Τέλος, στην τελευταία διαφάνεια προτείνω... Ναι. Προτείνω το εξής ε, κάποιους τρόπους που ακριβώς εξετάζουν αυτές τις προοπτικές. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να κατονομάζουμε την παιδική φτώχεια και να έχουμε έναν στόχο που θα αφορά τα παιδιά. Όπως ξέρετε έχουμε έναν γενικό στόχο 20 εκατομμυρίων αλλά δεν το έχουμε καθορίσει. Πρέπει να το καθορίσουμε γύρω από τα παιδιά και αν θέλουμε να περιλάβουμε και την εγγύηση για τα παιδιά προτείνω να στοχεύσουμε το 2,5% των παιδιών εκείνων που έχουν και τους τρεις όρους αυτούς ε, στον ορισμό του ΙΡΟΠ, δηλαδή που ζουν σε νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας, σε νοικοκυριά με σοβαρές ηλικέ ελλείψεις ε, και χαμηλής έντασης εργασίας. Ε, αλλιώς μπορούμε να εργαστούμε βάση το χάσμα αυτό της φτώχειας Επίσης προτείνω και γίνεται ήδη πάρα πολλή δουλειά επ' αυτού ότι η επίτευξη του στόχου θα πρέπει να μπαίνει στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και γενικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στις συστάσεις ανά χώρα και θεωρώ ότι το σχέδιο ψηφίσματος του Απριλίου σημείωσε μεγάλη πρόοδος προς αυτό. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να δουν αυτήν την ιδέα και στο ψήφισμα και στις ιδέες Κομισιόν όπου υπάρχει ιδέα ενός προϋπολογισμού για τα παιδιά, συγκεκριμένων μέτρων για τα φτωχά παιδιά, κινήτρων επίσης και τέλος πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η εγγύηση για τα παιδιά είναι πολύ περίπλοκη και άρα μάλλον δεν θα μπορέσει να εισαχθεί στους πέντε αυτούς τομείς ε, βράχει πρόθεσμα, οπότε θα πρέπει να επιλέξουμε μια ακολουθία. Ε, πιθανώς ε, δε ο πιο σημαντικό τομέα να είναι η προσχολική φροντίδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Υπήρξατε πολύ συγκεκριμένοι. Εσείς έχετε το λόγο, τα μέλη της Επιτροπής μας, για ερωτήσεις, τυχόν σχόλια. Κύριος Πάτων. Ευχαριστώ. Είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα για όλους μας στο μέλλον. Τα σχόλιά σας είναι άκρως ενθαρρυντικά. Όσον αφορά την ε, προσέγγιση που ακολουθείτε, τους στόχους που έχουν τεθεί και τη δέσμευση που έχει αναλυφθεί. Έχω κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω αν είναι σωστές για αυτή την Επιτροπή. Εγώ τι θέσω όμως. Η πρώτη. Τι με ενδιαφέρει τα αποτελέσματα του εγχειρήματο. Στην παρουσίαση αναγνωρίσατε τα θέματα, τα προβλήματα, την κλίμακά τους. Παρουσιάσατε συστηματική προσέγγιση στα προβλήματα. Τα αποτελέσματα όμως να βγουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους από τη φτώχεια. Είναι περίπλοκο. Πώς γίνεται. Χρειάζεται πολύ χρόνο και ίσως διαφορετική αξιολόγηση και προσμέτρηση των επιτευγμάτων. Θεωρία της αλλαγής θα μπορούσα να αποκαλέσω. Δεύτερον, εγώ μακρόν ασχολήθηκα με το θέμα στην πράξη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα από τα προβλήματα που είχαμε, κυρίως χρησιμοποιώντας τους πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιο ήταν – η περιπλοκότητα και η γραφειοκρατία κυρίως για μικρούς ε, φορείς και οργανισμούς να έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη. Κυρίως στην περίπτωση της φτώχειας των παιδιών, πολύ συχνά η χρηματοδότηση και τα προγράμματα πάνω στους συνήθους υπόπτους μεγάλους φορείς, κοινότητες, οργανώσεις, φιλανθρωπικούς οργανισμούς, διότι έχουν δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την ατέρμονα διαδικασία υποβολής αλλά δεν είναι όμως αναγκαία οι που εργάζονται στην πρώτη γραμμή και έρχονται σε άμεση επαφή με τους νέου που αναφέρατε και το πείσατε. Αυτή η πρωτοβουλία που επικροτώ για να είναι επιτυχής, θα είναι επιτυχής εάν βρούμε τα χρήματα που θα διατεθούν σε εκείνους που μάχονται στην πρώτη γραμμή. Η κυρία Ροβόλσκα. Całkiem niedawno Ευχαριστώ. Η αυτοματοποίηση, η οικονομία, η πράσινη, ε, η αγορά εργασία. Αναφερθήκαμε σε αυτά πριν. Τώρα μιλάμε για τη φτώχεια των παιδιών. Πρέπει δημοσία να πούμε ένα πράγμα. Είναι πολύ θλιβερό, διότι επί σειρά ετών μιλάμε για την φτώχεια των παιδιών με στις πολυμελείς οικογένειες που παραμένουν αδρανείς στο περιθώριο. Λέμε ότι οι αρμοδιότητες είναι στα χέρια των 100 μελών. Να πω τι γίνεται στην Πολωνία. Το 2016 ξεκίνησε το πρόγραμμα 500 συν για τις οικογένειες. Έτσι απεκλήθη αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που μείωσε τη φτώχεια των παιδιών και στην Πολωνία βρήκαμε, βρήκαμε ότι υπήρξε μείωση πράγματι της στόχες των παιδιών. Η πιο μεγάλη πτώση σε αυτό το στοιχείο από την πτώση του κομμουνισμού. Κατά την άποψή μου, σε κάποιες χώρες λείπει η επαρκής αποφασιστικότητα για τη μείωση της στόχιας των παιδιών. Λένε ότι δεν υπάρχει επαρκής ανάπτυξη σε κάποιες χώρες, ότι η αγορά εργασίας δεν είναι ευνοϊκή. Και είναι ντροπή να χρησιμοποιούν αυτά τα επιχειρήματα. Να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και να εξακολουθούμε να έχουμε το πρόβλημα. Όταν δρομολογήσαμε αυτό το πρόγραμμα στην Πολωνία φοβόμασταν ότι οι γυναίκες θα σταματούσαν να εργάζονται, ότι ότι θα αυξανόταν παθολογικές συμπεριφορές όπως ο αλκοολισμός. Αντίθετα, δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Οι οικογένειες ε, συμπεριφέρθηκαν υπεύθυνα και εκτιμούν και προσπαθούν να διατηρήσουν τις καλές συνθήκες για τα παιδιά τους. Η πολιτική των κρατών μελών πρέπει να δώσουν τα σωστά κίνητρα για να ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος. Η κυρία που μας έκανε την παρουσίαση αναφέρθηκε σε προσεγγίσεις βάσει των υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, των υπηαγωγείων κλπ. Ενίσχυση που χορηγείται στις οικογένειες, οικονομική. Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση κατά την άποψή μου και όχι τομεακή. Εν τη αυτή περίπτωση, κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει η παιδεία ο εκπαιδευτικός τομέας. Έχω μία ερώτηση. Πώς βλέπετε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για τη στήριξη της οικογένειας στα κράτη-μέλη. Μπορούμε να πούμε αν μπορεί να μειωθεί η φτώχεια των παιδιών χωρίς να μιλήσουμε για πολιτική για τις οικογένειες χωρίς να αναφερθούμε στο δεσμό που υπάρχει, ή τη διασύνδεση που υπάρχει με την οικογένεια. Δηλαδή, χρειάζονται πολιτικές επαρκείς για τις οικογένειες, εάν δεν είναι καλές οι πολιτικές της οικογένειας, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια των παιδιών ακολουθούν. Δεν θα εξαφανιστούν. Ευχαριστώ κυρία Ραφάλτσκα. Ήταν τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που θέλετε να θέσετε. Όχι. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τέλη για να απαντήσει στις τεθήσεις ερωτήσεις. Ε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από τη τελευταία ερώτηση. Να επιτρέψετε να πω ότι συμφωνώ μαζί σας σε κάποιο βαθμό ότι υπήρξε ανεπαρκής δραστηριότητα όσον αφορά τη φτώχεια των παιδιών και πολλά κράτη-μέλη δεν κάνουν επαρκείς προσπάθειες. Εγώ είμαι κοινωνιολόγος και αυτό που με εκπλήσει είναι η αναγνώριση των παιδιών σαν άτομα αυτά κάθε αυτά και που έχουν δικαιώματα. Αυτό είναι τεράστιο ταξίδι για πολλές κοινωνίες για να γίνει. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα παιδιά ή μάλλον δεν τα βλέπουμε καν τα παιδιά από πολλές πλευρές. Πρέπει να κάνουμε αυτό το ταξίδι, να αλλάξουμε, να σκεφτούμε τα παιδιά σαν άτομα. Και αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα που προέβαλα. Να πούμε ότι πρέπει να τα δούμε ατομικά δεν σημαίνει ότι τα βγάζουμε από την οικογένεια ή δεν σκεφτόμαστε ότι είναι ενταγμένα σε ένα πλαίσιο οικογενειακό και βέβαια πρέπει να τα θεωρήσουμε στο οικογενειακό πλαίσιο. Έχετε δίκιο λοιπόν. Πράγματι, η ενίσχυση της οικογένειας οδηγεί σε ενίσχυση των παιδιών από πολλές πλευρές, κυρίως στήριξη σε μετρητά. Διαφορετικά τα πράγματα βέβαια με τις υπηρεσίες και σχετικά με την φροντίδα των παιδιών σε μικρή ηλικία, νηπιαγωγία κλπ. Αυτό είναι κάτι που συνήθως αφορά τους γονείς και όχι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Τι προτείνω εγώ να βάλουμε, να προβάλλουμε στην πρώτη γραμμή τα παιδιά όσο γίνεται, αλλά να μην τα απομονώσουμε από τους γονείς, να μην θεωρήσουμε ότι η ευημερία τους είναι διαφορετική από αυτή των γονέων. Τουλάχιστον να έχουμε σαν άμεσο στόχο τα παιδιά και μετά εάν έχουμε σαν συγκεκριμένο στόχο τα φτωχά παιδιά. Δεν είμαι απεσιόδοξη. Υπάρχει κάποια αλλαγή να θεωρηθούν τα παιδιά ως άτομα Υπάρχει προβληματισμό για την ευημερία το οποίο διαβίωση των παιδιών από πολλέ πλευρέ. Εγώ τα βλέπω κάπω πιο αισιόδοξα από ότι εσεί. Ξέρω το πρόγραμμα το πολωνικό το 500 συν είχε σημαντικό αντίκτυπο στον αφορά τη μείωση τη φτώχεια και τη οικογένειακή φτώχεια. Σας ευχαριστώ για αυτή την παρατήρηση. Τώρα για τα αποτελέσματα. Την άλλη ερώτηση. Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα στόχο, ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, να εξαλείψουμε την πολυδιάστατη φτώχεια από το 2,5% πληθυσμού, δηλαδή περίπου 2,5 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη. Αυτό είχα υπόψη μου, σαν ενδεχόμενο στόχο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Εξαιρετικά δύσκολος πληθυσμός αυτός, διότι εκεί έχεις ανθρώπους που πιθανότατα είναι οι πιο στερημένοι. Αν αυτό όμως είναι το πνεύμα της εγγύησης, μπορούμε να προβάλλουμε ένα επιχείρημα για να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι δυσχερέστατο να βρούμε την επιτόπια χρηματοδότηση μέσω των παρόντων θεσμών, κυρίως ε, όσον αφορά τους μικρούς φορείς σε τοπική κοινότητα κλπ. Δεν έχω μαγικό ραβδί για κάτι τέτοιο. Συμφωνώ μαζί σας, δίκιο έχετε για αυτό που λέτε και σας ευχαριστώ. Απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Να καλωσορίσω τους, το νέο μας φιλοξενούμενο, τον κύριο Χόγκαρτ, Τέρενς Χόγκαρτ, Νατσιόνε Τζάκομο Προλίνη, Φοντατσιόνε Τζάκομο Προλίνη, αυτό μπορώ να πω. Καλώς ήρθατε και έχετε το λόγο για να μας κάνετε την παρουσίαση σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να έρθουμε εδώ. Μεγάλη χαρά για μένα. Τι θα ήθελα να πω. Θα ανακαλύψω κάποια από τα στοιχεία που ήδη εξατέθησαν σε πρώτερες παρουσιάσεις του ILO και του ΟΣΑ και ίσως εδώ ακολουθούμε παρόμοια προσέγγιση. Θέλω να αναφερθώ στην πολιτική για τις και το ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης και της σχετικής πολιτικής και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Διάφορες αρνητικές αλλαγές ίσως να είναι στον ορίζοντα. Πώς θα αντιμετωπιστούν από πλευράς Ευρώπης και πολιτών της μέσω δεξιοτήτων και μέσων προσαρμογής. να πούμε εξ αρχής ότι είχαμε πολλά επιτεύγματα όσον αφορά τη βελτίωση των δεξιοτήτων στην Ευρώπη τα τελευταία 10-20 χρόνια. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Τα προβλήματα που μας περιμένουν δεν έχουν εύκολες λύσεις. Και κάποια προβλήματα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αύξηση δεξιοτήτων, εκμάθηση, αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι μακρά διαρκείας. Αλλά υπάρχουν σημάδια ότι έχουν πετύχει βελτιώσει κάποιε τομεί. Να πω λοιπόν ευθύ εξ αρχής ότι ζητάμε πολλά από την πολιτική δεξιοτήτων. Σε επίπεδο 100 μελών διαβάσατε τα κατάλληλα έγγραφα. Βλέπετε ότι βελτιώνουμε το επίπεδο του ανθρωπίνου κεφαλαίου και λέμε ότι θα τα πάντα. Γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί, έτσι λένε στα κάτι μελη είναι πιο ικανοποιημένη η κοινωνία, πιο χαρούμενη, επενδύσουμε σε δεξιότητε. Στην πραγματικότητα, οι δεξιότητε είναι ένα κομμάτι πακέτου μέτρων. Σημαντικό στοιχείο, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα. Για να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση καλέ, να βελτιώσουμε τι συνθήκε αν θέλουμε ευρωπαϊκή οικονομία με υψηλέ δεξιότητε και υψηλέ αμοιβέ. Οι δεξιότητε παίζουν ένα ρόλο, αλλά δεν είναι ο μόνο παράγον. Δεν μπορούμε να το δούμε κάτι, σαν κάτι απομονωμένο. Να διατρέξω κάποια βασικά στοιχεία, βασικέ τάσει που διαβλέπουμε στο μέλλον. Συζητήθηκαν το πρωί. Τεχνολογική αλλαγή, με άλλα λόγια. Ε, παγκοσμιοποίηση πράσινη οικονομία, δημογραφική αλλαγή. Σημαντικέ προκλήσει αυτό που είναι αρκετά ενδιαφέρον είναι τα εγκάρσια θέματα. Πρόσφατα, τι είδαμε. Τεχνολογικές αλλαγές. Δημιουργήθηκαν κενά έτσι στην αγορά εργασίας. Κάποιες θέσεις με υψηλές δεξιότητες προωθούνται. Και κάτω, στο κάτω επίπεδο, σε εργασίες χαμηλών δεξιοτήτων. Αύξηση. Στο μέσο έχουμε κάποια κενά και εξαφανίσεις θέσεων. Και όπως προαναφέρθηκε υπάρχει και πόλωση της απασχόλησης. Καλές θέσεις εργασίας και κακές. Κάποιες κακές δουλειές μπορεί να είναι πολύ κακές. Αν αντιμετωπίζει ο κόσμος την κατάσταση που δεν ξέρει ότι μία μέρα στην άλλη αν έχει δουλειά. Και δεν είναι σίγουροι ότι θα έχουν εισόδημα τη μία μέρα στην άλλη αν θα βγάλει το κάματο. Μη τυπικές μορφές εργασίας, αν εργάζονται σε πλατφόρμες κλπ. Είναι πραγματικό πρόβλημα αυτό. Και κάτι άλλο που παρατηρείται. Έγιναν σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Άρα ο κόσμος έχει πιο πολλά προσόντα και δεξιότητες. Παράλληλα, βλέπουμε πρόβλημα να ταιριάσουν οι δεξιότητες με τις ανάγκες. Οι επενδύσεις που έγιναν με άλλα λόγια σε ανθρώπινο κεφάλαιο δεν αποπληρώνονται, δεν δίνουν αποτελέσματα για κάποιους που βρήκαν δουλειά που δεν χρησιμοποιεί, δεν χρησιμοποιεί τις δεξιότητές τους. Και είδαμε σε έρευνα ότι 25% του εργατικού δυναμικού λέει ότι τα προσόντα τους δεν ταιριάζουν στη δουλειά που κάνουν. θεωρούν ότι έχουν παραπάνω προσόντα για τη θέση τους ή λιγότερα. Και απειρχαιωμένες δεξιότητες υπάρχουν. 47% των θέσεων εργασίων στην ΣΥΠΑ μπορούν να αντικατασταθούν φερρυπίν, έτσι λέγεται, από αυτοματοποίηση. Αυτά είναι αποτελέσματα που βγαίνουν στους τίτλους. Ο ΣΑ δείχνει 14% σε αυτό και ΣΕΝΤΕΦΟΠ ε, έχει κάνει έρευνες και δείχνει ότι 8% ε, θέσεων απασχόλησης ε, που μπορεί να θεωρούνται σαν πεπαλαιωμένες και να χαθούν λόγω αυτοματοποίησης. Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι είναι παρόλα αυτά. Και αν είσαι ένας από αυτά τα 2 εκατομμύρια είναι πρόβλημα. Έχουμε δύο διαγράμματα. Βλέπουμε τις παρελθούσες αλλαγές και το πώ έχει αλλάξει η αγορά εργασία και δημιουργήθηκαν κενά, στο άλλο διάγραμμα βλέπετε μελλοντική αλλαγή. Προβλέψει του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Τι βλέπουμε. Πού θα, βρούμε, πού θα υπάρχουν οι δουλειές στο μέλλον. Τι είναι ενδιαφέρον. Υπάρχουν απαιτήσει για την κατάσταση. Πολύ μεγάλες απαιτήσει. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας Κάποιε θέσει δεν μπορούμε να τις διαβλέψουμε σήμερα, να τι προβλέψουμε. Θα απαιτούνται νέε δεξιότητες. Την επόμενη δεκαετία περισσότερη αλλαγή θα είναι απλή κανονική, όπου οι φυστάμενες δουλειές θα βγουν στη σύνταξη κάποιοι, ας πούμε, και θα πρέπει να καλυφθούν οι θέσεις των συνταξιούχων. Και αυτές οι θέσεις μπορεί να αλλάξουν, αλλά θα αλλάξουν πιθανότατα λίγο, όχι πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που λένε το μέλλον, ότι γρήγορα θα αλλάξουν τα πάντα και θα εξαφανιστούν αύριο κάποιες θέσει θέσεις εργασίας, δεν είναι κάτι που θα συμβεί απαραίτητα. Στην πραγματικότητα η αλλαγή ε, γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς. Εγώ ξεκίνησα την εποχή που γινόταν επανάσταση με τους μικροεπισεργαστές και ακούγαμε ιστορίες τρόμου τότε. Αλλά η τεχνολογία τελικά, όπως είδαμε, είναι υποφελής. Um, if we just look at uh, um, what's been happening over the recent Να δούμε τι έγινε στο πρόσφατο παρελθόν. Υπάρχουν και καλά μαντάτα στην Ευρώπη. Είδαμε ότι αυξήθηκαν οι δεξιότητες και τα προσόντα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση και τα σχετικά συστήματα πλησίασαν περισσότερο τις ανάγκες αγοράς εργασίας. Υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση αναγκών προσόντων. Η προσέγγιση εδράζεται επί των αποτελεσμάτων. Τα τελευταία 20 χρόνια περίπου είδαμε η επαγγελματική κατάρτιση και η παιδεία να έγινε το βασικό μονοπάτι που ακολουθείται σε κάθε κράτος μέλος. Για τους νέους έχει γίνει μια επιλογή και είναι αποτελεσματικός τρόπος για μετάβαση προς την αγορά εργασίας. Αν δείτε τους στόχους για το 2020, υπάρχουν πολλά στοιχεία ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος. Για εκείνους που φεύγουν νωρίς από το εκπαιδευτικό σύστημα, να, οι ενήλικες να συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και να μπαίνουν περισσότεροι νέοι στην ε, ανώτατη παιδεία. Έχουμε και καλά, καλές εξελίξεις. I'm clearly failing the technology aptitude test here. go. Okay, so that's it, challenges. Challenges? Okay, now it's right. Okay. Yeah, so, um, so the, the, the, but there are a major set of... Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις και προβλήματα. Πολλά από αυτά είναι μακροχρόνια προβλήματα η επαγγελματική κατάρτιση και η παιδεία μπορεί να είναι αποτελεσματική. Το δείχνει η έρευνα του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Η απόδοση για του νέου που περνάνε από επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση μπορεί να είναι πιο υψηλή από ότι για μεγαλύτερη ηλικία. Α, μάλλον από ότι να μπει κανείς κανονικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά δεν θεωρείται ω πρώτη επιλογή η επαγγελματική κατάρτιση. Κάνουμε διάκριση μεταξύ αρχική επαγγελματική κατάρτιση, όπω μαθητεία κλπ, και απόκτηση δεξιοτήτων και κατάρτιση των ενηλίκων, των πιο μεγάλων. Τα θεωρούν σαν κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Γιατί οι πιο μεγάλοι να μην έχουν πρόσβαση σε πολλέ δραστηριότητε κατάρτισης που εντάσσονται στην αρχική φάση. Η διαβίω εκμάθηση παραμένει ένα πρόβλημα για πολλέ ευάλωτε ομάδε, ηλικιωμένα άτομα και πιο περιθωριακές ομάδες αγοράς εργασία πολύ συχνά για τον εργοδότη δεν συμφέρει να κάνουν την επένδυση. Και η αγορά από μόνη της δεν θα λύσει αυτά τα προβλήματα. Και πώς αντιμετωπίζουμε την το να είναι πεπαλαιωμένες οι δεξιότητες όταν οι άνθρωποι είναι ακόμα στη δουλειά τους αντί να περιμένουμε να χάσουν τη δουλειά τους πρώτα. Και το πρόβλημα των βασικών δεξιοτήτων είναι ένα πρόβλημα και αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αρκετά δραστηρία, ιδιαίτερα δραστηρία όσον αφορά την πολιτική τις δεξιότητες. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει. Μπορούμε να εντοπίσουμε όμως κάποια παρόμοια θέματα. Βελτίωση πρόσβαση για κάποιες ομάδες στην κατάρτιση. Και από πλευράς κοινωνικής συνοχής τα βλέπουμε αυτά. πώ βελτιώνουμε την ποιότητα τη κατάρτιση που χορηγείται και πώς αξιολογούμε τη δεξιότητα των ανθρώπων, κυρίως αν έχουν αποκτηθεί μέσω επίσημης και ανεπίσημης κατάτησης και πώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Και διάφορες πολιτικές πώς συμβάλλουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανθρώπων. Και για να πετύχουμε μια Ευρώπη που επιθυμούν οι πολιτικοί. Χρειάζεται βελτίωση συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την αγορά εργασία. Ο Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ε, το θεματολόγιο για τι δεξιότητε είναι πολύ σημαντικό. Το δικαίωμα των ανθρώπων στην ε, πρόσβαση στι δεξιότητε και στην κατάρτιση και η ατζέντα για τι δεξιότητε θέλει να βελτιώσει τι δεξιότητε, να βελτιώσει τον αριθμό ανθρώπων που έχει δεξιότητε, να υπάρχει τέριασμα προσφορά ζήτηση και να γίνεται σωστή εξακρίβωση των δεξιοτήτων. Πέραν αυτών, Έχουμε μαθητεία, ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις μαθητείες, ευρωπαϊκή συμμαχία για τη μαθητεία που προώθησε την εκμάθηση, κάτι πολύ επαντασματικό, εβδομάδα για τις δεξιότητες επαγγελματικέ και την κατάρτιση, έτσι ο κόσμος να θεωρεί ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι πρώτη επιλογή. Έγιναν πολλές επενδύσεις από το Κοινωνικό Ταμείο πάνω σε αυτά. Υπάρχει επίσης το διάφορα προγράμματα για να βελτιώσουμε τα διάφορα συστήματα, να μαθαίνει το ένα κάτω μέλο από το άλλο και το, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Κατάρτιση και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ έκανε ανάλυση και έρευνα για να μάθουμε από τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, να κατανοήσουμε α, το τι είναι αποτελεσματικό. Έχουμε Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση που, που εξετάζει το πλαίσιο, πώς μπορεί να βελτιωθεί για να καλυφθούν πολλά προβλήματα που αναφέραμε όσον αφορά την πολιτική δεξιοτήτων και για τα επόμενα χρόνια και για την εκμάθηση των ε, μεγαλυτέρων. Έχουμε το ψήφισμα του Συμβουλίου για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, για την εκμάθηση δεξιοτήτων από τους ενήλικες, τη διαβίω εκμάθηση, την ανάγκη να μάθει κανείς να είναι ευέλικτο, να μην υπάρχουν αδιέξοδα, ποιοι παρέχουν την εκπαίδευση αυτή, να υπάρχει σωστή ποιότητα και το θέμα της χρηματοδότησης. Πώς θα χρηματοδοτείς όλα αυτά. Κυρίως όταν η απόδοση της επένδυσης, η απόσβεση της επένδυσης είναι προβληματική όσον αφορά κάποια άτομα. Αν οι εργοδότες επενδύουν. Η πλατφόρμα για τον, ε, να ανταλλάσσονται γνώσεις κλπ. και η ατζέντα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο δεξιοτήτων των ατόμων, όπου αυτά οι δεξιότητες λείπουν να υπάρξει μια κινητικότητα, άνοθη κινητικότητα. Όλα αυτά ήταν υποφελή μέτρα τα τελευταία 10-20 χρόνια. Βελτίωσαν το, πολιτι... το, το τον των πολιτικών όσον αφορά τις δεξιότητες, την επαγγελματική κατάρτιση κλπ. Το μέλλον. Τι γίνεται, ποια είναι τα βασικά θέματα. Υπάρχουν επίμονα θέματα δύσκολα να την αντιμετωπίσει. Στο μέλλον, η επαγγελματική εκπαίδευση σημαίνει ότι χρειάζεται μια ευρεία βάση να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα με άλλα λόγια. Διάφοροι φορεί τη αγορά εργασία, όπω κοινωνικοί εταίροι, πρέπει να βοηθήσουν το σχεδιασμό. Ξέρουν τις ανάγκες της αγοράς, πρέπει να συμμετάσχουν το IVET για τους ενήλικες, για τους μεγάλους, πρέπει να προωθηθεί. Η μαθητεία ε, μπορεί να δώσει νέες δεξιότητες ακόμα και σε μεγάλους ανθρώπους. Χρειάζεται κατάθεση σε όλα επίπεδα, να υπάρχουν αδιέξοδα. Να μπορείς να μεταπηδάς από επίπεδο σε επίπεδο. Αναβάθμιση δεξιοτήτων. Ο καθένας με κάποιο τρόπο να μπορεί να έχει το δικαίωμα απόκτησης δεξιοτήτων με αποτελεσματικό τρόπο. Άρα χρειάζεται προσανατολισμός. Χρειάζεται βελτίωση προσανατολισμός των ενηλίκων. Άρα, έλεγχος των τεκτενωμένων στην αγορά εργασίας. Για να γίνονται επενδύσεις που θα σχετίζονται με την τρέχουσα και μελλοντική ζήτηση. Να μην γίνονται επενδύσεις που πάνε στράφη. Αυτό που κάνει σε ΔΕΦΟΠ είναι σημαντικό στην Ευρώπη. Και εκτό Ευρώπη τι γίνεται. Και ο σάμποια μπορεί συμβάλλει. Με προσανατολισμού. Εν συντομία λοιπόν, αυτά πρέπει να συμβούν στο μέλλον και ευχαριστώ. Thank you for the presentation. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Υπάρχουν ερωτήσεις, μάλιστα. Μια ερώτηση. Laro, you, the floor is yours, and then, oh, sorry, Mr. Goiken is next, and behind him, Mr. Betten. Betten. Τρεις ερωτήσεις έχουμε. Παρακαλώ εσείς πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Πισλάρου. Είναι η δεύτερη παρουσίαση που ακούσαμε μετά το που το Σεντεφόπ και πραγματικά είναι ευχάριστο να ακούμε και είναι καλό που βλέπουμε ότι μεταξύ σας ε, ε, συνεργάζεστε για να έχετε μια ε, πλήρη εικόνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ε, και το γεγονός ότι πρέπει να αναπτυχθεί αυτό, αυτό το είδους η επαγγελματική κατάρτιση έχουμε δυσκολίες όσον αφορά τις ε, δεξιότητες που χρειάζονται. Ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν πως είναι επαγγελματική κατάρτιση ε, συμπλήρωμα για αυτούς που δεν είναι αρκετά ταλαντούχοι και αυτό είναι εις βάρος ε, του σωστού επίπεδου εκπαίδευσης που θα πρέπει να προσφέρεται. Υπάρχουν επίσης διαφορετικές ε, απόψεις. Εγώ προέρχομαι από τη Ρουμανία όπου βασικά το όριο ήταν ότι οι, φοιτητές, οι, μαθητές που δεν έμπαιναν πάνω από πέντε αυτόματα πηγαίνανε προς την επαγγελματική παιδεία. Αυτό όμως αποτελούσε στίγμα για τα παιδιά αυτά και, σημαίνει, και σήμαινε ότι ε, εντάξει, αφού δεν, δεν μπορείς να διαβάσεις, ε, άντε να γίνεις υδραυλικός. Ότι ένας υδραυλικός δεν έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα να, να διαβάσει το Στογεύσκι, ας πούμε. Ε, ε, εμείς πώς μπορούμε να διευρύνουμε αυτή την αντίληψη, πώς να ενσωματώσουμε την, ενσωματώσουμε την παιδεία, την καλλιέργεια με την ε, επαγγελματική κατάρτιση και παιδίου. Βλέπουμε ότι θα πρέπει να συνδυαστεί η μη τυπική ε, κατάρτιση. Μιλώντας μόνο για επίσημη επαγγελματική κατάρτιση και παιδεία, ξεχνάμε τις μαθητείες και τα Δεν θέλω να αμφισβητήσω το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, δεν ήταν ε, και άλλωστε πρέπον, αλλά εσείς ε, τι έχετε να μας συμβουλέψετε εδώ εμάς τους νομοθέτες. And Mr. Äh, αυτά τα οποία μας είπατε. Θα ήθελα να πω πως οπωσδήποτε η ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας θα δημιουργήσει προβλήματα. Βεβαίως θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Το σημαντικό για εμένα είναι να εστιάζουμε στους ανθρώπους γιατί βλέπουμε ότι αυξάνεται πάρα πολύ ο ρυθμός εργασίας και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να ανταποκριθούν και φεύγουν από τον κόσμο εργασίας γιατί καταραίουν. Αυξάνεται πάρα πολύ αυτός ο αριθμός από χρόνο σε χρόνο. Πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την ψηφιοποίηση με το να δημιουργήσουμε κάποιο πλαίσιο έτσι ώστε ο κόσμος να μην καταραίει υπό το βάρος όλης αυτής της διαβίου κατάρτισης. Εξάλλου τι νόημα έχει αν δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί και τον αρρωσταίνει ο χώρος εργασίας. Κάτι άλλο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται δύο ή και τρεις δουλειές για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα επίπεδο ζωής. Και ακριβώς εδώ πέρα ε, τίθεται το ζήτημα. Με συγχωρείτε, αν θα μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο αργά για να σας ε, καταλάβουν και οι διερμηνείς. Λοιπόν, εντάξει, θα μιλήσω λίγο πιο αργά. Όπως είπα, χρειάζεται ο ε, κόσμος να κάνει δύο-τρεις δουλειές για να μπορέσει να διατηρήσει ένα επίπεδο ζωής και εδώ πέρα ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα της οικογένειας. Αν αρρωστήσει ο μπαμπάς ή η μαμά και φεύγει από τη δουλειά, ε, είναι προγραμματισμένο πλέον ότι θα έχουμε μια, κοινωνική κατάπτωση και βλέπουμε ότι αυξάνεται πολύ γρήγορα και παιδική φτώχεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λοιπόν, και δημιουργούνται πλέον αιστείε κοινωνική ένταση στην Ευρώπη που πλέον κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να αντεχθούν. Έχετε σκεφτεί να απευθυνθεί ο κανονισμός αυτός για το χώρο εργασίας στους ανθρώπους και όχι στην ψηφιοποίηση. Γιατί ε, μας λέτε εδώ πέρα, ε, πράγματι μπορεί να αποτελέσει η ψηφιοποίηση μια ευλογία με το να μειώσει τον ρυθμό εργασίας. Χοντρικά αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστούμε κύριε Γκόικινγκ. Ο κύριος Πάτεν έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω διάφορα σχόλια και ερωτήσεις. Ωραία, συγγνώμη. Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω. Εγώ χαίρομαι που ακούω ότι η κατάσταση εδώ πέρα βελτιώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί όλα τα στατιστικά στοιχεία που βλέπω εγώ λένε ότι η κατάσταση εξαρτάται κατά πολύ από την κάθε περιοχή. Ίσως να βελτιώνεται ο μέσος όρος, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία αυτό δεν συμβαίνει. Μιλάμε για την παιδική φτώχεια πάντα έτσι. Δεύτερον, θα συμφωνούσαμε με τα σχόλια που έγιναν στην πρώτη ερώτηση. Έχουμε την εντύπωση πως υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις ε, κουλτούρας, αν θέλετε, στην επαγγελματική κατάρτιση σε σχέση με παραδοσιακή ακαδημαϊκή οδό και μέχρι να το δούμε αυτό πάντα θα αποτελεί ένα ζήτημα. Δεν δέχομαι αυτό το οποίο είπατε για τα συμβόλαια μηδενικών ορών τα οποία απορρίπτεται. Εγώ θα έλεγα ότι για πολλούς ανθρώπους αυτά τα συμβόλαια είτε είναι φοιτητέ, είτε εργαζόμενοι γονείς είναι κάτι το πάρα πολύ χρήσιμο γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δημοφιλές. Δεν διαφωνώ ότι κάποιοι εργοδότες ε, τα χρησιμοποιούν, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει και αναπτύσσεται και δεν πρέπει να το αγνοούμε. Η ε, πραγματική μου ερώτηση αφορά κάτι το συγκεκριμένο και αφορά την φτώχεια στον χώρο εργασίας. Οπωσδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε μια αύξησή του τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως η αύξηση των δεξιοτήτων φαίνεται θεωρητικά να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αλλά υπάρχουν πραγματικά προβλήματα συχνά ε, σε νοικοκυριά όπου και οι δύο ενήλικες ε, εργάζονται και το να αναλάβουν ε, τέτοια εκπαίδευση όπως φαίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι κάτι το οποίο είναι ακριβό οικονομικά και από πλευράς χρόνου θα πρότεινα πέρα από το να σκεφτούμε το πώς θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν δεξιότητες που χρειάζονται για την αγορά, να σκεφτούμε και δομικά πώς θα δομηθεί η επαγγελματική κατάρτιση, καθώς να θα πρέπει να μπορέσει να έχει πρόσβαση η συγκεκριμένη ομάδα που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Ευχαριστώ. Κυρία Μπίσοφ ε, έχει τον λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Θα ήθελα να γνωρίζω το εξής μιλάμε για τις προκλήσεις, το τι προκαλεί τις αλλαγές. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν την δυνατότητα στους ανθρώπους να καταρτιστούν καλύτερα. Έχετε κάποιες προτάσεις για το πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Έχουμε τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και εγγυάται ε, όχι μόνο στον καθένα το δικαίωμα στην εκπαίδευση, αλλά, διαβάζω από μέσα, ε, ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλισμούς, ε, διαβίου εκπαίδευση και την δυνατότητα να διαχειριστεί καλύτερα τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Να δούμε λοιπόν πώς οι δρόντες ή αυτοί οι οποίοι είναι συλλογικέ διαπραγματεύσεις ή τα κράτη θα μπορούσαν να υλοποιήσουν αυτά τα δικαιώματα των πολιτών. Αλλιώ ε, θα, θα φαίνεται σαν μια ατομική πρόκληση. Ε, Βεβαίω δεν ήμουν εδώ πέρα στην αρχή γιατί ήμουν και στην Επιτροπή Οικονομικών για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την Κοινωνική Διάσταση. Πού βλέπετε εδώ πέρα τις ε, πρόπτικες αυτού του ζητήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, τελευταία ερώτηση ή μου ξέφυγε κάποιος όχι. Κύριε Χόγκαρτ, μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση. Έχετε τον λόγο. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Να ξεκινήσω με την τέταρτη ερώτηση. Να ξεκινήσω το τέλος. Ε, λέει η πολιτική ότι ο κόσμος πρέπει να έχει δικαίωμα, αλλά πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Υπάρχει περιθώριο να δούμε βεβαίως ε, την πλευρά των ατόμων, ε, των κοινωνικών εταίρων, το πώς θα μπορέσουν να εγγυηθούν κάποια δικαιώματα. Ειλικρινά όμως δεν ξέρω ποια θα είναι η απάντηση. Ε, πρέπει όμως να έχουν τα άτομα τη ε, δυνατότητα. Δηλαδή εύκολα μπορεί να λέμε έχει κάποιο δικαίωμα, αλλά αν δεν μπορούν να το ασκήσουν, να το υλοποιήσουν, ε, δεν έχει νόημα. Πρέπει να βρεθεί κάποιο τρόπο να μπορέσουν να το υλοποιήσουν και νομίζω τα καλύτερα τα οποία έχουμε είναι συλλογικέ συμβάσει και κοινωνικέ συμβάσει οι οποίε θα δίνουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε κατάρτιση και θα δώσουν και την ε, δυνατότητα σε κόσμο που είναι εκτός του κόσμου της εργασίας να μπει, αλλά πρέπει να υπάρχει και πάρα πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση για το τι ε, χρειάζεται να μάθει κανείς. Δηλαδή, εάν επιδοτήσουμε απλά την κατάρτιση με κάποιον τρόπο, ε, έχουμε μια κατάρτιση για την κατάρτιση, χωρίς να ανταποκρίνεται σε κάποια πραγματική ανάγκη της αγοράς. σε σχέση με την πρώτη και τρίτη ερώτηση. Ναι, εντάξει, σωστό αυτό το οποίο είπατε για την οικονομία με τις πλατφόρμες, αλλά ε, γεγονό είναι ότι υπάρχουν και πολύ κακές δουλειές ε. αλλά γεγονό είναι ότι αυτοί που κάνουν αυτές τις δουλειές δεν έχουν εύκολα πρόσβαση σε κατάρτιση. Το θεμελιώδες ε, ζήτημα είναι το πώς ξεπερνάμε αυτήν την διάκριση μεταξύ γενικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι ένα ακαθόδες ζήτημα, δηλαδή ως ένα βαθμό είναι μια τεχνητή διάκριση την οποία μπορούμε να ξεφορτωθούμε. Δηλαδή πολλά τέτοια προγράμματα πλέον, τα παραδοσιακά προγράμματα εκπαίδευσης πλέον κοιτάνε την απασχολησιμότητα. Και είναι κατ' ουσίαν προγράμματα επαγγελματική κατάρτισης, απλά ε, με άλλο όνομα. Οπότε είναι μια τεχνητή διάκριση. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να το δούμε μακροπρόθεσμα για να ξεπεράσουμε αυτό τον διαχωρισμό. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε μέσω πρόθεσμα είναι να δείξουμε ότι αυτός ο τρόπος τους επιτρέπει να ενταχθούν και στην ανώτατη εκπαίδευση. Γιατί αυτός είναι ένας παράγοντας που νομίζει ότι ε, είναι κάτι το δεύτερο, γιατί δεν θα μπορέσω να πάω σε ένα πανεπιστήμιο εάν ακολουθήσω αυτήν την πορεία. Λοιπόν, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να το δουν αυτό και να το κάνουν, να ανοίξουν και οι πύλες από εκεί. Λοιπόν, αν υπάρχει μια καλή ιστορία, αν θέλετε, για τις ανταμοιβέ που έχει α, αυτή η σταδιοδρομία. Γιατί καμιά φορά επικρατούν λάθος αντιλήψεις για την αξία της επαγγελματικής κατάρτισης και αυτό θα είναι θετικό. Στη δεύτερη ερώτηση για την ποιότητα της εργασίας. Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε αργότερα, αλλά νομίζω ότι επανέρχεται σε αυτό το οποίο είπαμε πριν ότι δηλαδή ζητάμε πάρα πολλά από την πολιτική δεξιοτήτων και η ικανότητα ας πούμε, να ανταποκριθεί στο το οτι ότι κάποιος έχει δύο-τρεις δουλειές ε, είναι λίγο υπερβολικό να το ζητάμε. Είναι αρμοδιότητα άλλων τομέων. Λοιπόν, αυτά και ζητώ συγγνώμη αν δεν απάντησα πλήρως είναι ζητήματα περίπλοκα. Υπάρχουν εδώ και 20-30 χρόνια και θα συνεχιστούν. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα τα κάνουμε καλύτερα. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση που ήρθατε και που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Πάμε τώρα παρακάτω σε έναν άλλο καλεσμένο. Καλωσορίζουμε τον Φρανκ Χέντριξ από το Καθολικό Πανεπιστημίο της ε, Λέβεν. Καλώς ήρθατε. Έχετε τον λόγο. Παρακαλώ, ξεκινήστε. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ε, όλα τα μέλη της Επιτροπής που μου καλέσατε σήμερα εδώ. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το νομικό πλαίσιο το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το εργατικό δίκαιο και την οδηγία για την απασχόληση. Ε, θα αναφερθώ από, στις βασικές αναφορές και ζητήματα που προκύπτουν όταν κανείς μιλά για ε, εργασιακό δίκαιο και ε, δίκαιο απασχόλησης. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να πούμε ότι αν μιλάμε για εργατικό δίκαιο στην Ευρώπη, βασικά μιλάμε για κάτι που ε, είναι πολύ καλά εδρεωμένο στα εθνικά συστήματα, στα κράτη-μέλη. Μας αποτελεί μέρος των παραδόσεων, των δομών των κρατών και του, της κουλτούρας των κρατών μελών και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη, απο, μεγάλη διαφοροποίηση στο εργατικό δίκαιο στην Ευρώπη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πρωτοβουλίες περί ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν έχουν πιστήσει προσοχή στις κοινωνικές πολιτικές και στην εργασιακή νομοθεσία στο παρελθόν με την υιοθέτηση του κοινωνικού κεφαλαίου το, στις αρχές του 90 και εφόσον έγιναν και κάποιες αναφορές ένα μεγάλο ε, σε, ορόσημο είναι ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό ο, νόμος για τα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν ξέρω αν βλέπετε καλά τώρα αυτή τη διαφάνεια αλλά το νομικό πλαίσιο συνδέεται όχι μόνο με τη συνθήκη και το κοινωνικό κεφάλαιο και αυτό θα λένε ανέκαθεν ναι, οι δικηγόροι ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δράσει θα πρέπει κάπως να αναφέρεται σε μια διάταξη της συνθήκης επί ε, από την οποία μάλλον απορρέει η αρμοδιότητά της να ενεργήσει. Άρα λοιπόν το κοινωνικό ε, κεφάλαιο τομέας ε, ε, αρμοδιότητας είναι σημαντικός, αλλά και οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να δούμε τους κανόνες ανταγωνισμού και τους κανόνες για την απασχόληση που υπάρχουν στη συνθήκη. Όταν μιλάμε, ας πούμε, για εσωτερική αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και εργαζομένων, αυτό έχει τεράστια επιρροή στα εργασιακά δικαιώματα. Παράδειγμα, η οδηγία απόσπασης εργαζόμενων. Εάν μιλήσουμε για ε, πολιτικές απασχόλησης, μιλάμε για ένα πλαίσιο συντονισμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη, τις πολιτικές τους και τις πρακτικές τους. Ίσως εκεί να μην είναι τόσο η νομοθεσία ο τρόπος να προχωρήσουμε, αλλά περισσότερο η ενημέρωση, η ανταλλαγή πρακτικών και οι κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη-μέλη για το μίσο που έχουν την πλήρη αρμοδιότητα. Ο ανταγωνισμός είναι ένας άλλος τομέας που ήθελα να αναφέρω, διότι έχουν υπάρξει θέματα ε, στον Ευρωπαϊκό Νόμο περί ανταγωνισμού, όταν αναφερόμαστε ας πούμε, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις ε, οι συμφωνίες οι συλλογικές έχουν συζητηθεί στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με βάση τους κανόνες ανταγωνισμού που λένε ότι οι ρυθμίσεις περί ε, συγκεκριμένων ε, τιμών ε, είναι αντίθετοι με τους κανόνες ανταγωνισμού. Βέβαια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επιτρέψει εξαίρεση ε, λέγοντας ότι λόγω των κοινωνικών στόχων των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις, σύμφωνα με τις παραδόσεις μας στην Ευρώπη οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες αντιτράστ και άρα θα πρέπει να επιτρέπονται σύμφωνα με το ε, νομοθεσία ανταγωνισμού. Όμως αυτές οι αποφάσεις περιορίζονται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τις εργατικές συνθήκες με πολύ παραδοσιακό ε, τρόπο και θα δούμε στο μέλλον Πώς αυτό θα θεωρηθεί όταν θα μιλάμε για συλλογικά συμπεφωνημένες ε, ε, συνθήκες για τους αυτοαπασχολούμενους στην αγορά εργασίας. Και θα επανέλθω σε αυτό. Τώρα, αν δούμε το κοινωνικό κεφάλαιο, που είναι η βάση για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στον τομέα της απασχόλησης, βλέπουμε ποια είναι η βάση για τον νομοθέτη του Ευρω... τον Ευρωπαίο και βλέπουμε το άρθρο 153 που έχει αποτελέσει βάση ας πούμε στο παρελθόν για την υγεία και ασφάλεια, το χρόνο απασχόλησης, την ίση μεταχείριση, την ευέλικτη εργασία, την προσωρινή εργασία, την ισορροπία ε, ανάμεσα στην οικογενειακή και την εργασιακή ζωή, ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους. Ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων έχει ήδη συμπεριληφθεί στις οδηγίες και θα βρείτε στο ενημερωτικό έναν κατάλογο των κυρίων οδηγιών που ισχύουν στον τομέα αυτό. Τώρα επίσης σας έχω υποδείξει ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους διάφορους τομείς όπου ισχύει η ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και τους τομείς όπου είναι πιο ευαίσθητοι και εκεί ε, ισχύει η ομοφωνία. Και εκεί θα δούμε πράγματα τα οποία ίσως στα συστήματα των κατών μελών ε, είναι πιο αμφισβητήσιμα, πιο συζητήσιμα ή πιο ε, ευαίσθητα. Μιλάμε για την προστασία της πάυσης της απασχόλησης, όταν δηλαδή μία σύμβαση λύεται. Μιλάμε για εκπροσώπηση των εργαζομένων και συλλογική άμυνα, ε, υπεράσπιση. Μιλάμε για εργαζόμενους τρίτων χωρών και για κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια. Θα δείτε όμως ότι όλα αυτά δεν αρκούν <clears throat> όσον αφορά την παραπομπή στο συνθήκη, στο νομικό πλαίσιο της συνθήκης, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για ορισμένους τομείς που αποκλείονται. Τομείς για τους οποίους η συνθήκη λέει πως αυτό δεν μπορεί να είναι υπόθεση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στόχους κοινωνικής πολιτικής. Και αυτό έχει να κάνει με τους μισθούς, το δικαίωμα της ε, οργάνωσης και το δικαίωμα της απεργίας. Ε, αν δούμε το θέμα των μισθών που αποκλείεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ξέρουμε ότι σε άλλου τομεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με, την, με τις αμοιβέ, γιατί όταν μιλάμε για την απόσπαση εργαζομένων υπάρχει μια διάταξη για ίσης, ίση αμοιβή, για τι ίσες ευκαιρίε, ίση αμοιβή για άνδρες και για γυναίκε. Α πούμε, και ένα σωρό αναφορέ άμεσε ή έμεσε στι αμοιβέ. Όμως εδώ είναι αυτό που συζητάτε για τη ρύθμιση ενός ε, ελάχιστου ευρωπαϊκού ημερομιστίου, ίσως αυτό να είναι παραβίαση της συνθήκης. Υπάρχουν προτάσεις από διάφορους θεσμούς να σκεφτούμε ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο ημερομίσθιο που θα βασίζεται σε ένα ποσοστό ενός μέσου όρου των εθνικών μισθών. Πάντως από νομικής άποψης αυτό θα είναι προβληματικό. Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες βέβαια έχει να κάνει με την πάυση μιας ε, σύμβασης εργασίας. Αναφέρθηκα σε αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, υπόκειται σε ομοφωνία. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον νομοθέτη ε, γιατί τα δικαιώματα αυτά θεωρήθηκαν ανέκαθεν θέματα των κρατών μελών. Αλλά είναι δυνατόν να γίνει κάτι σχετικά με αυτό από την ευρωπαϊκή άποψη, ε, προοπτική. Ακούγονται διάφορες φωνές ε, ε, από τους επαΐοντες ότι μπορούν να κάνουν κάτι ας πούμε για την ευελιξία, ε, και άρα έτσι να μιλήσουν και για δικαιώματα παύσης σε σύμβασης. Πάντως, από νομικής άποψης δεν θα είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Και δεν βλέπουμε μηνύματα εξάλλου να ασκείται καμία πίεση από τους πολιτικούς κύκλους για αυτά τα θέματα. Ένα άλλο σημείο που θέλω να θίξω είναι οι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Βλέπουμε ότι από τη μια πλευρά ε, λέει ότι η κοινωνική εταίρεια, ο κοινωνικός διάλογος ε, είναι παράδοση στις χώρες μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παίζουν και στρατηγικό ρόλο στην ε, χάραξη πολιτικών. Ο κοινωνικός χάρτης αλλά και ο πολιτικός, ε, ο χάρτης μάλλον αποφάσεων, ε, προβλέπει ε, ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα συμμετέχουν στην χάραξη πολιτικής, συνάπτουν ευρωπαϊκού εύρου συμφωνίες, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και άρα και η συσχέτιση αυτού του δικαιώματος με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις παραμένει μη ρυθμιζόμενος τομέας. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ευρωπαϊκών κανόνων και κανονισμών, παραμένει θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται με τις διεθνείς συμφωνίες, συλλογικές διαπραγματεύσεις, εφόσον δεν ρυθμίζονται από νόμο τότε δεν μπορούν να ρυθμίζονται από οποιοδήποτε νομικό σύστημα. Το θέμα είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ρόλο στην ρύθμιση των νομικών προϋποθέσεων ή όρων για να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για τη σύναψη συμφωνιών μετά από διεθνεί συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει και πάλι να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο κοινωνικό ε, χάρτη. Τώρα, ε, τέταρτη παρατήρηση σχετίζεται με νομικό θέμα, αλλά και με τα όσα αναφέρθηκαν σήμερα το πρωί. Ένα από τα θέματα λοιπόν είναι πώς ορίζουμε τον εργαζόμενο. Είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε ποιο είναι ο εργαζόμενος, γιατί τα δικαιώματα στη αγορά εργασία εξαρτώνται από το αν έχει καθεστώς εργαζόμενου και από νομική άποψη. Αυτό που βλέπουμε από νομική άποψη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει ένα νομιόμορφο αυτόνομο νομικό ορισμό του ποιο είναι ο εργαζόμενο. Έχουμε διάφορε έννοιε σε διάφορα σημεία της συνθήκης και σε διάφορα σημεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά δεν είναι μια ομοιόμορφη ευρωπαϊκή έννοια και συχνά ο Ευρωπαίος νομοθέτης παραπέμπει στην εθνική έννοια για να ορίσει το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών περί απασχόλησης. Άρα λοιπόν η εθνική νομοθεσία ορίζει πιο συνεργαζόμενος και άρα η ευρωπαϊκή νομοθεσία ισχύει για τον ευρωπαϊκό ορισμό του ποιο συνεργαζόμενος. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές στην εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσίας, σε ασάφεια και σε προβλήματα για τους αυτοαπασχολούμενου. Συσχετιζόμενο με την έννοια του εργαζόμενου είναι και το θέμα του για ποιον ρυθμίζουμε την αγορά εργασίας και για ποιον ρυθμίζουμε τις συνθήκες εργασίας. Εφόσον υπάρχουν νέες μορφές εργασίας, θα πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουμε με αυτές τις νέες μορφές, τι κάνουμε με τους αυτοπασχολούμενους. Και για το εργατικό δίκαιο το ίδιο είναι μεγάλη πρόκληση να σκεφτεί κανείς συνθήκες εργασίας για τους αυτοαπασχολούμενους. Αν δούμε τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά περιλαμβάνονται σε διάφορα διεθνή κείμενα, καταρχάς ο αυτοπασχολούμενος δεν αποκλείεται από μια ιδέα ότι δηλαδή είναι εργαζόμενος και άρα χρειάζεται να προστατεύεται. με όμως από τα εθνικά συστήματα ότι αυτά αντιμετωπίζουν τις κλασικές παραδοσιακές συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, ε, που τις έχουν διαπραγματευτεί μέσα από συλλογικέ διαπραγματεύσει, αλλά δεν προβλέπουν τίποτα για τους αυταπασχολούμενους. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευρύνει την αγορά εργασίας τους αυταπασχολούμενους. Άλλο ζήτημα είναι βέβαια οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους αυτοπασχολούμενους. Κάτι τέτοιο θα σημάνει ένταση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αντιτράστ και ελεύθερου ανταγωνισμού. Θα υπάρξει ένταση ανάμεσα στις συλλογικά συμπεφωνημένες συνθήκες για τους αυτοπασχολούμενους και τους κανόνες αντιτράστ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία το σημείο είναι η νέα τεχνολογία. Βλέπουμε ε, ότι υπάρχει συζήτηση για το εργατικό δίκαιο, για το γεγονός ότι ο κόσμος δουλεύει διαφορετικά, σε διαφορετικά πλαίσια. Ο χώρος εργασίας, η έδρα, ε, τα ωράρια, εφόσον ο χρόνος δεν έχει πλέον σημασία σε ορισμένα πλαίσια απασχόλησης και βλέπουμε και ζητήματα όσον αφορά την ρομποτοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν ρόλο <clears throat> στη συσχέτιση μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ που γίνεται στο χώρο εργασίας. Μπορεί κανείς να μιλήσει για ιδιωτική ζωή, για λήψη αποφάσεων, ποια είναι η ευθύνη στο χώρο εργασίας. Αυτά είναι ζητήματα για το μελλοντικό εργατικό δίκαιο, αλλά είναι και θέματα λαβές για προβληματισμό για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Τι ώρα είναι. Προτείνω να συνεχίσουμε με τον επόμενο φιλοξενούμενο. Και μετά από αυτό θα μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις και θα θέσουμε τις ερωτήσεις στον κύριο Χέντριξ και τον κύριο Καμπρέλη και τον κύριο Καβλή. I see no nose Everyone Is agree so. Let's do that. Αν συμφωνείτε, καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο. Uh, Στην Επιτροπή μας, Υγεία και Ασφάλεια στον τόπο εργασίας του μέλλοντος είναι ο τίτλος. Έχετε το λόγο. Thank Πρόεδρε, και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Τιμή για μένα να έρθω να σας μιλήσω και προνόμιο είναι κοινή παρουσίαση. Ο καθηγητής Χέντριξ και εγώ θα μιλήσουμε. Είμαι και εγώ νομικός και ο Dr. Richard Graveling από το Ινστιτούτο Ιατρικής Εργασίας είναι ειδικό όσον αφορά την ε, ασφάλεια στον τόπο εργασίας και την υγεία. Θα μιλήσουμε για πολιτικές στον τόπο εργασίας του μέλλοντος και αυτό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχετικού Νόμου. Η παρουσίασή μου έχει τέσσερα τμήματα. Μια εισαγωγή που παρουσιάζω τις διάφορες τεχνολογίες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τόπο εργασίας και ποιες είναι νέες μορφές οργάνωσης του περιβάλλοντος εργασίας που δημιουργούν αυτές οι νέες τεχνολογίες, οι αρνητικές και εντοπίζω ενδεχόμενους κινδύνους και πραγματικούς κινδύνους όσον αφορά την υγιεινή ασφάλεια που είναι απόρρια των νέων τεχνολογιών και των νέων τρόπων εργασίας. Ενδεχόμενες και πραγματικές. Τονίζω τους δύο αυτούς όρους. Διότι για κάποιες μορφές εργασίας οι κίνδυνοι ήδη φύστανται. Ο καθηγητής Χέντριξ αναφέρθηκε προηγουμένως σε κάτι στο πεδίο που καλύπτει η έννοια εργαζόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ενωσιακό δίκαιο. Και μετά θα αναφερθώ σε ενδεχόμενους κινδύνους και τι κενά υπάρχουν στην υφιστάμενη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ε, νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σώμα νομολογίας, χωρίς να θέλω να κάνω λογοπαίγνια, που είναι υγιή. Έχουμε 24 ευρωπαϊκέ οδηγίε και την οδηγία για το χρόνο εργασίας που είναι κάπως ξεχωριστή. 25 οδηγίες που μπαίνουν σε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την υγεία και ασφάλεια. Και στο τέλος θα συναγάγω συμπεράσματα. Πάμε στο πρώτο τμήμα. Εισαγωγή. Μου ζητήθηκε να αναφερθώ σε κάποιες αρνητικές τεχνολογίες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο, γι' αυτό είναι αρνητικές, στο περιβάλλον εργασίας. Κυρίως η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση και η χρήση των ρομπότ στον τόπο εργασία. AR και VR, η τεχνητή ε, πραγματικότητα, η εικονική πραγματικότητα και αυξημένη πραγματικότητα, VR και AR. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτούς τους όρους. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι οι αλγόριθμοι στη ροή των εργασιών. Έχετε αναθέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ένα πιλωτικό πρόγραμμα περί αλγορίθμων και πώς οι αλγόριθμοι επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων, όχι μόνο στο περιβάλλον εργασίας, αλλά εν γέννη. Πέρα από την έξω στην ευρωπαϊκή κοινωνία, για τους σκοπούς της παρουσιάσεως, να πω το εξή. Οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται από κάποιους εργοδότες και χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να παρακολουθούν το προσωπικό, αλλά για να διαχειρίζονται τις επιδόσεις και να προβλέψουν και την αντίδρασή τους, τη συμπεριφορά τους σε κάποια προβλήματα στον τόπο εργασία, πώς θα τα αποκριθούν, σε κάποια ενδεχόμενα, πώς θα τα αποκριθούν. Όλα αυτά για προώθηση και αύξηση της παραγωγικότητας χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο, όχι απλώς για εποπτεία και παρακολούθηση. Εποπτεία και παρακολούθηση είναι ένα κομμάτι του ρόλου τους, αλλά και προβλέψει πραγματικό χρόνο της συμπεριφοράς και πώς αντιδρά ο κόσμος σε διάφορα που συμβαίνουν στον τόπο εργασίας. Π.χ. αλλαγέ. Έχουμε αυξανόμενο φαινόμενο άλλο. Το γνωρίζει καλά ο συνάδελφός μου. Η ψυχοφυσιολογία, οι εργοδότες χρησιμοποιούν τεχνικές παρακολούθησης για να προσμετρήσουν εγκεφαλικά, ε, ε, συμπεριφορά του εγκεφάλου, ένταση, οξυγόνωση και όλα αυτά για την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα. Όλες αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να είναι πολύ παρεμβατικές. Και ερχόμαστε λοιπόν έτσι σε ενδεχόμενους κινδύνους που δημιουργούν για την υγεία και ασφάλεια. Θα αναφερθώ σε αυτά αργότερα. Η προηγούμενη διαφάνεια αφορούσε τις τεχνολογικές αλλαγές. Μιλήσαμε και για την οικονομία σε, γι... γιγάντια κλίμακα που χρησιμοποιείται η τεχνολογία σαν ένα μέλος, σαν ένα τμήμα για νέες μορφές εργασίας. στον Αμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία ενδεχομένω και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είμαι σίγουρος έχουμε μηδέν ώρες. Οι, οι συμβάσει μη εγκυμένων ελάχιστων ωρών συμβάσεις για επιδόσεις που δεν εγγυώνται ώρες εργασίας. Ad ρύθμιση. Ο εργοδότης προσφέρει εργασία χωρίς δεσμεύσεις. Ούτε και το άτομο είναι υποχρεωμένο να δεχτεί εργασία αν ποτέ του προσφερθεί. Ένα τμήμα της ευρύτερης τάσεως. Ψευτοαπασχόληση. Αυτό που ανέφερε ο καθηγητής Χέντριξ και άλλοι η ψεύτο αυτοαπασχόληση, μηδέν ώρες ή συμβάσεις με μηδενικές ώρες εργασίες, γιγαοικονομία, πλατφόρμες εργασίας, δημιουργούν τα ίδια θέματα της κάλυψης. Ποιος καλύπτεται εντός του προστατευτικού μανδύα του εργασιακού δικαίου και υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια. που οι λεπτομέρειες αναφέρονται περισσότερο στο έγγραφο. Δεν μπορώ να αναφερθώ εκτενώς λόγω χρονικής πίεσης. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα. Δεύτερον τμήμα. Ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι και ενδεχόμενοι κίνδυνοι, θεωρητικοί κίνδυνοι. Το πρώτο που πρέπει να υπογραμμίσω είναι ότι υπάρχει μέτριο επίπεδο έρευνας που έχει διεξαχθεί μέχρι τώρα. Αυτό που διαθέτουμε είναι κάποια στοιχεία περί ψυχοκοινωνικών βλαβών και κινδύνων που σχετίζονται με τη νέα Αυτό που θεωρεί ότι είσαι πάντα διαθέσιμο εργοδότη. Με αναμένω το τηλέφωνό σου, πάντα θα είσαι έτοιμο να ανταποκριθεί στι ανάγκε του πελάτη και τη δουλειά. Όποτε απαιτεί η υπηρεσία ο εργοδότη σου. Είναι ψυχοκοινωνικέ βλάβε λόγω Επίσης, αν κανείς είναι βαπτισμένος σε εικονική πραγματικότητα, δημιουργεί βλάβες. Έχουμε κάποια στοιχεία για ψυχοκοινωνικές βλάβες που προέρχονται από την γίγα οικονομία, αυτοαπασχόληση, συμβάσεις μηδενικών ωρών και εργασία εξ αποστάσεως. Έχουμε κάποια στοιχεία για αμυοσκελετικές διαταραχές. Και αυτό στα πλαίσια κοινών αυτοματοποιημένων τόπων εργασίας. Δηλαδή, εκεί που οι άνθρωποι και τα ρομπότ ε, έχονται σε επαφή μεταξύ τους. Κάποιο αυτόματο μηχάνημα, ένα ρομπότ, παράγει κάποια δραστηριότητα και ένας άνθρωπος απαιτείται να είναι δίπλα ή να αλληλεπιδρά με το μηχάνημα ή το ρομπότ και κάποια φορά, κάποιες φορές αυτό οδηγεί σε μυσκελετικές διαταραχές και προβλήματα. Όμως αυτά τα στοιχεία είναι σποραδικά ατελή και γι' αυτό στις επόμενες διαφάνειες, όπου έχω κάποιο πίνακα που αναφέρεται σε ενδεχόμενους και πραγματικούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια, εντόμισα τις ψυχοσωματικές βλάβες, μειοσκελετικές διαταραχές και δυνατότητα φυσικών συγκρούσεων μεταξύ ρομπότ ή αυτόματων συσκευών και ανθρώπων. Είναι μια δυνατότητα. Τι λέω. Άρα λέω ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω έρευνα πάνω σε αυτά πληρέστερη ανάλυση αυτών που συμβαίνουν. Όπως βλέπετε, από τον πίνακα έχω εντοπίσει κάποιους πραγματικούς κινδύνους για την υγεία και ασφαλεία. Σε ψεύτο αυτοαπασχόληση, συμβάσεις μηδενικών ορών, οφείλονται αυτά, τεράστια οικονομία, γιγαοικονομία και εργασία σε πλατφόρμες και αυτό αφορά τον ορισμό του εργαζομένου στα πλαίσια του εργασικού δικαίου. Ο εργαζόμενος είναι ο άξονας επί των οποίων οι κανόνες περιγές και ασφάλειας βασίζονται. Αν δεν είσαι εργαζόμενος δεν έχει δικαίωμα στην υγεία και ασφάλεια. Και οι ευθύνε που πέφτουν στα πλαίσια της ε, νομοθεσίας, της κείμενης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να εξασφαλίσετε ότι ο χώρος εργασίας είναι υγιεινός και ασφαλής και περιβάλλον είναι κάτι ασαφές σχετικά με αυτό. Αυτό τι σημαίνει. Ότι αυτό που έχουμε είναι νομοθετικό κενό. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που παρέχουν προσωπική υπηρεσία που δεν καλύπτονται από το σχετικό δίκαιο περί υγείας και ασφάλειας. Γιατί, θα με ρωτήσετε, γιατί κάποια άτομα που είναι σε κεκαλυμμένη αποσχόληση, είναι στην γίγα οικονομία, συμμετέχουν σε εργασία, σε πλατφόρμα ή αποστάσεως εργασία, γιατί δεν θεωρούνται εργαζόμενοι. Χρειάζεται να παρέχεται μια προσωπική υπηρεσία, βλέπετε. Και η νομική ανάλυση ποια θα ήταν. Αν αυτά τα άτομα μπορούν να σε επαφή με πολλούς ενδεχόμενους πελάτες, δεν υπάρχει αποκλειστικότητα παροχής υπηρεσίας. Δεν υπάρχει ένας φορέας προς τον οποίο να απευθύνεται η υπηρεσία υπάρχει πάνω από έναν εργοδότη εντό εισαγωγικών. Το εργοδότη εντό εισαγωγικών. Και αυτέ οι πολλέ μορφέ εργασία σημαίνει η δυνατότητα που έχει το άτομο να αντικαταστήσει να αντικατασταθεί από κάποιον άλλον και να παράσει την υπηρεσία. Άρα δεν είναι προσωπική υπηρεσία αφού μπορεί να αντικατασταθεί αυτό που παρέχει την υπηρεσία από κάποιον άλλον συνάδελφο. Και δεν θεωρείται εργαζόμενο με αυτόν τον τρόπο, με την έννοια τη νομοθεσία. Αν πήγα πίσω, ζητώ συγγνώμη. Ποια είναι τα κενά. Αν υποθέσουμε ότι αυτοί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι υπάρχουν. Έχουμε στοιχεία, κάποια στοιχεία και θεωρούμε ότι μπορεί να είναι και πραγματική κίνδυνη. Τι κάνουμε. Έχουμε την εξής κατάσταση. Ίσως θέλουμε να εξετάσουμε μια νέα οδηγία για, χημικά και φυσι... για χημικούς και φυσικούς κινδύνους να περάσει. 24 οδηγίες, οι σχετικές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποδιαιρούνται σε 5 γενικές οδηγίες, 3 οδηγίες για τύπο εργαζομένου που αφορούν μερική απασχόληση, φερρυπίν και άλλα διεργασίες, 5 το... με συγκεκριμένο τομέα που καλύπτουν, ορυχεία, ε... σκάφη, ε, πλοία, και οδηγίες για φυσικούς κινδύνους που καλύπτουν συγκεκριμένους κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια, σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα ήταν λογικό λοιπόν να εντοπιστεί ότι υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί για φυσικούς κινδύνους, ψυχοκοινωνικούς κινδύνους μια οδηγία. Λιγότερη ριζική πρόταση θα ήταν όμως οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που προέρχονται από την αυτοματοποίηση, ψεύτο αυτοαπασχόληση και όλα αυτά ανακαλύπτονται στα πλαίσια γενικής αναθεώρησης, περιοδικής αναθεώρησης των κειμένων νομοθεσιών, των σχετικών. Που το κάνετε συχνά. Το βασικό κενό, ενδεχομένως, αφορά τους ψυχοκοινωνικούς ε, κινδύνους και την πνευματική υγεία, την ψυχική υγεία. Υπάρχουν και άλλοι ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Σχετίζονται με μειοσκελετικά προβλήματα. Επαναλάβω όμως ότι η κείμενη νομοθεσία έχει κενό. Διότι πολλά από αυτά τα άτομα στην ψεύτο αυτοαποσχόληση και γίγα οικονομία Κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, αλλά σημαντικό ποσοστό τους, δεν θεωρούνται εργαζόμενοι, άρα δεν καλύπτονται από βασικούς κανόνες και πρότυπα περί και ασφάλειας στον τόπο εργασίας. Άλλα νομοθετικά προβλήματα είναι οι μυοσκελετικές διαταραχές και οι κίνδυνοι να δημιουργηθούν αυτές οι διαταραχές επανειλημμένα έχει αναφερθεί σε έρευνες όσον αφορά την κινημένη νομοθεσία περί και ασφάλειας. Και μόνο κάποιες οδηγίες καλύπτουν αυτές τις διαταραχές. Και άλλα και να υπάρχουν ίσως όσον αφορά τις πράσινες τεχνολογίες και εναλλακτικέ ενεργειακές πηγές και την αλλαγή των πρακτικών στην εργασία που περιστρέφεται γύρω από την πράσινη τεχνολογία, Φερρυπίν. Αλλαγές στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και νανοηλικά κλπ. Και υπάρχει και κενό όσον αφορά την νομοθεσία περί καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων. Όσον αφορά τα νανοηλικά και τα νανομόρια. Εν κατακλείδη. Όπως σας είπα υπάρχουν κάποια στοιχεία όσον αφορά ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, μυοσκελετικές διαταραχές, αυτοματισμός, ρομποτική αλγόριθμοι, ψεύτο αυταπασχόληση κλπ. Μερικά στοιχεία. Δεν υπάρχει πλήρη κάλυψη και δεν είναι εμπεριστατωμένα τα στοιχεία. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Πρέπει να ανατεθεί. Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, τότε αυτό συνεπάγεται ενδεχομένως τροποποίηση της κείμενης σχετικής νομοθεσίας. Να θεσπιστούν να θεσπιστεί μια οδηγία για φυσικούς κινδύνους ή αυτοί οι κίνδυνοι να ενταχθούν εντός μιας αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Κύριε Γκράβελινγκ, θέλετε να προσθέσετε κάτι ίσως. Όχι θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Ε, ωραία, σας ευχαριστώ. Έχετε λοιπόν τον λόγο. Εσείς ε, οι βουλευτές ε, της Επιτροπής θέλετε να κάνετε κάποιες προτάσεις, παρατηρήσεις. Κυρία Μπέσα, Μπίσοφ. Έχω να κάνω μια παρατήρηση. Δεν σας προξένησε έκπληξη, γιατί ακούσαμε τι προκλήσεις έχουμε στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής πως ε, δεν αναφέρεται καθόλου ο τομέας αυτός στην επιστολή της υποψήφιας επιτρόπου. Παρακαλώ. Είναι ενδιαφέρον ας πούμε. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Ναι. θεωρείται ε, θέμα στο οποίο υπάρχουν διαφωνίες κυρίως επειδή ε, δεν ε, είναι πια τόσο σαφής διάκριση μεταξύ δουλειάς και αναψυχής και λοιπόν δραστηριοτήτων ακούσαμε κάποιον να λέει ακριβώ το πώς υπάρχει αυτό το πράγμα στον τομέα της υγείας εγώ αύριο είμαι σε ένα εργαστήριο για μειοσκελετικές διαταραχές και την πρόληψη τους που τα έχουμε εδώ και 30 χρόνια και δεν έχει το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις ε, για αυτό το κομμάτι της ε, συζήτησής μας. Όχι, εάν δεν υπάρχουν... Ναι, να κάνω άλλο ένα σχόλιο. Μιλήσαμε για την αλλαγή του ορισμού του εργαζόμενου και τα κενά στον ορισμό. Κάτι το οποίο δεν αναφέραμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο χώρος εργασίας. Η νομοθεσία είναι 25-30 ετών και μιλήσαμε ε, για το ότι συνεχώς μιλάμε για παραδοσιακή εργασία. Εσείς κάθεστε εδώ πέρα, τα απόγευμα δουλεύετε, χρησιμοποιείτε υπολογιστές κάποιου είδους. Ποιος είναι υπεύθυνο για τον χώρο εργασίας σας για τις καρέκλες στις οποίες ε, κάθεστε που δεν πάνε στο κατάλληλο ύψος στα προβλήματα για τον λαιμό σας ε, εάν συνέχεια σκύβετε και κοιτάτε την ταμπλέτα ε, αυτό εδώ είναι χώρος εργασίας δεν καλύπτεται όμως από τον κανονισμό περιοφωνών Δηλαδή η ιδέα αυτή του ότι αλλάζει η αντίληψη του χώρου εργασίας, μιλήσαμε για την ισορροπία ζωής και εργασίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Δηλαδή, εάν είναι κατάλληλη πλέον η νομοθεσία. Ευχαριστώ. Επειδή έπρεπε να φύγω νωρίς, δεν είχα την ευκαιρία να κάνω ερωτήσεις προς την ε, κυρία Νταλή για την εγγύηση για τα παιδιά και οφείλω να πω πως Ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε κονδύλια, έργα, προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας, ειδικά της παιδικής. Και παραδείγματο χάρη εγώ είμαι από την Σλοβακία. Και εκεί πέρα είχαμε τα κονδύλια για να χρησιμοποιήσουμε για τους Ρωμά που επηρεάζονται πάρα πολύ από τον κίνδυνο φτώχειας εκεί τα παιδιά. Και τα χρησιμοποιήσαμε, κάναμε τα έργα ε, και δεν άλλαξε τίποτα. Ε, οι αριθμοί χειροτέρεψαν, οπότε όταν μιλάμε για το θέμα της παιδικής φτώχειας, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά αυτή τη φορά, έτσι ώστε τα λεφτά να χρησιμοποιηθούν με τρόπο αποτελεσματικό. Σας ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση. Κοιτάξτε, η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχει εδώ πέρα μια δυναμική, δηλαδή μαθαίνουμε όσον αφορά την παιδική φτώχεια. Νομίζω ότι είναι ακόμα κάτι το οποίο είναι καινούριο ως πολιτική. Έχουμε πολιτική καταπολέμησης της ε, φτώχειας ε, όσο έχουμε ε, φτώχεια, αλλά δεν το έχουμε δει από την σκοπιά των παιδιών και με καθέ σεβασμό θεωρώ πως οι πολιτικές των Ρωμά επίσης είναι γενικές πολιτικές σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα αυτή και η αίσθησή μου είναι ότι με την εγγύηση υπάρχει η δυνατότητα να ορίσουμε τα παιδιά ως δικαιούχους των επιδομάτων ε, δεν είναι τόσο κοινό αυτό και δεν έχει συμβεί και ήδη ε, εσείς αν μπορώ να πω και η ε, Κομισιόν ε, είναι κάπου εκεί ε, όσον αφορά τον καθορισμό των στόχων, το να κατονομάζει παιδιά ως ομάδα προτεραιότητας είναι κάτι το καινούριο, δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής εξ όσων γνωρίζω στο πολιετές πλαίσιο 2014-2020 δεν αναφέρονταν συγκεκριμένα τα παιδιά τώρα υπάρχει μια πρόταση να αναφερθούν ότι οι συνθήκες όπου τα κράτη-μέλη πλέον θα έχουν στρατηγικές κατά της φτώχειας οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία τα οποία αφορούν τα παιδιά και τις άλλες αρνητικές συνθήκες. Υπάρχει η πρόταση ενός δίκτυ παρακολούθησης που θα κατονομάζει τα παιδιά. Ήταν ε, μια ομάδα που είχε έναν δίκτυ, αλλά ίσως να είναι κάτι ευρύτερο από το FED και να μην πάει από το ε, τα 0 έως 15, αλλά 0 έως 18 οπότε τρόπον να ήδη έχετε κάνει αρκετά η πρόκληση θα είναι στις διαπραγματεύσεις που έρχονται να παραμείνουν και να διατηρηθεί το επίπεδο αυτό αν θέλετε αυτό το οποίο έχει προτείνει το κοινοβούλιο οπότε έχω την αίσθηση ότι ο καθορισμός ε, κονδυλίων σύνδεση με, τους, ε, με τις συστάσεις αναχώρα ε, η στόχευση των παιδιών ειδικά που δεν αναφέρονται βεβαίως δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο λοιπόν εάν γίνει η σύνδεση και με κάποιον τρόπο μπουν τα παιδιά στο επίκεντρο, χωρίς να αποκλείουμε τους ενήλικες ή άλλους, αλλά αν επικεντρωθούμε στα παιδιά, νομίζω έχουμε μια πολύ ισχυρή ιδέα που πρέπει να την σκεφτούμε. Ναι, οπωσδήποτε. Μια ερώτηση ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για παιδιά που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και να προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα. Αναφέρατε ας πούμε την εκπαίδευση, την προσχολική. Συμφωνώ, αλλά η κατάσταση διαφέρει τόσο πολύ από το ένα κράτος στο άλλο και τα παιδιά εκείνα τα οποία είναι κοινωνικά υστερούν ε, είναι εκτός ε, παιδικών σταθμών και αυτό ισχύει ειδικά στα κράτη-μέλη που έχουν ε, μια μεγάλη κοινοτάρωμα, ειδικά εκεί όπου ζει σε ξεχωριστούς καταβλισμούς. Οπότε αναρωτιέμαι αν έχετε τα δεδομένα. Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά αυτά τα οποία κινδυνεύουν από την φτώχεια. Ποια είναι η καλύτερη ηλικία. Κοιτάξτε, τώρα θεωρούμε ότι η καλύτερη ηλικία είναι μεταξύ 2 και 3 ετών μια πάρα πολύ σημαντική ηλικία για τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε μια έκθεση για το πώς εμφανίζονται τα παιδιά στο σχολείο και υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι κάποια πάνε με πάνες 4-5 ετών ότι δεν μπορούν να συντάξουν μια πλήρη πρόταση, δεν ξέρουν τι είναι ένα βιβλίο. Φαντάζομαι θα συμβαίνουν αυτά και σε άλλες χώρες αλλά η αίσθησή μου αυτή τη στιγμή είναι 2-3 ετών η κρίσιμη ηλικία και είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας γιατί αυτό το οποίο μαθαίνουμε ακόμα και σε χώρες με ε, υψηλή τέτοια παροχή τέτοιων υπηρεσιών είναι ότι υπάρχει ανισότητα και τα παιδιά δεν πηγαίνουν εκεί ε, και είναι αυτά τα οποία το χρειάζονται περισσότερο οπότε η ιδέα αυτή της ανισότητας Μιλάμε για την ποιότητα, μιλήσαμε για υπηρεσίες που θα πρέπει να είναι πρόσιτες, αλλά πρέπει να δούμε το θέμα της ανισότητας και τα στοιχεία τώρα α, ε, έρχονται ακόμα και όταν είναι δωρεάν μία υπηρεσία ή προσιτή. Τα φτωχότερα παιδιά δεν πάνε. Είναι και θέμα κουλτούρας. Ναι, ναι, συγγνώμη και είναι η τελευταία μου ερώτηση. Ξέρετε, εγώ είχα εργαστεί με τέτοια παιδιά και την κοινότητα των Ρώμα και για πολύ καιρό νομίζαμε ότι για να σπάσει ο φάβλος κύκλος θα έπρεπε να εστιάσουμε στην εκπαίδευση, αλλά οι βέλτιστες πρακτικές μας δείχνουν ότι είναι η στέγαση. Γιατί ακόμα και όταν τα σχολεία είναι δωρεάν δεν πάνε στα σχολεία γιατί ζουν σε τέτοιες ε, κακές ε, συνθήκες ώστε οι γονείς δεν ξυπνάνε το πρωί να τα πάνε στο σχολείο. Δεν τα ξυπνάνε τα παιδιά. Ε, είναι πολύ απλό δηλαδή. Είναι πολύ απλός ο λόγος για τον οποίο δεν πάνε σχολείο. Και αναρωτιέμαι αν με την εκπαίδευση στην προσχολική θεωρείτε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση των παιδιών να το κάναμε υποχρεωτικό. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας και βεβαίω ε, εκτός Ευρώπης, ειδικά στη Λατινική Αμερική και σε κάποια μέρη της Αφρικής, ε, έχουν ε, όρους για να δώσουν τα λεφτά στις οικογένειες, συχνά στις μητέρες μάλιστα, και τα παίρνουν τα λεφτά μόνο εάν το παιδί πάει σε μια κλινική ή σε κάποιο σχολείο και είναι θετικά τα αποτελέσματα. Η αίσθησή μου είναι ότι πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί γιατί συχνά έτσι κατηγορούμε τους γονείς και ειδικά τις μητέρες. Οπότε μπορεί να το σκεφτούμε αυτό, αλλά όχι από μόνο του. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα κίνητρα για τις οικογένειες, νομίζω, για να φέρουν τα παιδιά τους. Και η εκπαίδευση, όπως λέτε, είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίως ε, τώρα έχουμε προγράμματα που εκπαιδεύουν τους γονείς για την σημασία και να στηρίξουν επίσης τους γονείς, όχι να τους υπαγορεύουν, αλλά να προσπαθούν να αντιληφθούν την κατάστασή τους, γιατί γονείς που δεν μπορούν να σηκωθούν το πρωί από το κρεβάτι είναι σε μια κατάσταση ε, στέρησης και αυτή, όπως και αν το πούμε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, για το ότι ήρθατε εδώ και μοιραστήκατε αυτές τις πληροφορίες ε, μαζί μας και ελπίζω να παραμείνουμε σε επαφή γιατί έχετε τα δεδομένα, εμείς έχουμε τόσες ερωτήσεις ε, και τόσα άλλα ζητήματα να συζητήσουμε, οπότε μένουμε την συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ